Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε ακόμα περιορισμένος κύκλος, αλλά παρόλα αυτά θα αρχίσουμε. Διότι βεβαίως ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και ήδη αμέσως προσέρχονται δύο σημαντικοί προσκεκλημένοι. Γνωρίζετε ότι θα προσέλθει όσον ούπο ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι και αργότερα ο Πρόεδρος Μάιστατ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ας μη σπαταλούμε χρόνο, λοιπόν, έχετε την ημερήσια διάταξη, υποθέτω ότι δεν έχετε ενστάσεις. Να σας πω λίγο για την οργάνωση των εργασιών σήμερα, την οποία γνωρίζετε, αλλά θα το επαναλάβω. Ο εισηγητής μας θα κάνει εισαγωγή 5 λεπτών στο θέμα, μετά θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο για 10 λεπτά για την πρώτη του παρέμβαση και θα ακολουθήσουν για 4 λεπτά το πολύ ο καθένας οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και μετά θα προχωρήσουμε στη γενική συζήτηση. Θα γίνει ίσως και ένας γύρος πάλι απαντήσεων με τον Επίτροπο και τον ίδιο μηχανισμό θα ακολουθήσουμε και για τη συζήτηση με τον πρόεδρο Μάιστατ. Είναι λοιπόν σαφές ότι πρέπει όλοι να είμαστε πειθαρχημένοι, βεβαίως όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και όλοι όσοι θα λάβουν το λόγο σήμερα για τις ανακοινώσεις της Προέδρου τώρα, στις ανακοινώσεις της Προέδρου μάλλον, θα πω ακόμη ότι αν θέλετε ίσως κάνουμε και μια σύντομη ε, έκθεση σχετικά, την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή και μετά από πρόσκληση της Ουγγρικής Βουλής και ειδικότερα του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών της Ουγγρικής Βουλής βρέθηκα στη Βουδαπέστη μαζί ήταν και πολλοί άλλοι πρόεδροι συναρμόδιων επιτροπών των βουλών των χωρών μελών είχε λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον ο ευρύς αυτός κύκλος έμαθα πολλά πράγματα έτσι νομίζω για το πώς συζητούν οι βουλές των χωρών μελών την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Στην δε δική μας των προϋπολογισμών θα έχουμε την ευκαιρία τον Απρίλη να συζητήσουμε με βουλευτές των Εθνικών Βουλών. Προσπάθησα βέβαια επίσης, πιστέψτε με, και το έπραξα και το τόνισα κατ' επανάληψη, ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένουμε τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή, να είναι παρά το πλευρό μας, να είναι σύμμαχοί μας και όχι αντίπαλοι μας. Είμαστε φυσικοί σύμμαχοι, εν μέρη μάλιστα και αντιμέτωποι με, τις, με ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις. Ορισμένοι συμφώνησαν και εν τέλει παρόλε τις αρχικές μου επιφυλάξεις διεπίστωσα ότι ήταν χρήσιμη η επαφή αυτή. Άλλη ανακοίνωση. Ορισμένοι που παρακολουθούν διαρκώς την ιστοσελίδα μας θα το έχετε διαπιστώσει. Υπάρχει τώρα πάντως το έγγραφο εργασίας υπαριθμών 3 που περιλαμβάνει τα, τα πορίσματα στα οποία έχουμε καταλήξει στην συζήτησή μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τώρα στην ιστοσελίδα μας όλα τα έγγραφα πλήρως. Είπαμε επίσης ότι η επόμενη συνεδρίασή μας η οποία θα γίνει στο Στρασβούργο, είναι παρένθετη αυτή, θα ασχοληθεί με δύο θέματα. Αφενός με την ευρωπαϊκή υπηκότητα και αφετέρου με την αλλαγή του κλίματος. Η Επίτροπος Χέντεγκάρτ ανακοίνωσε ωστόσο ότι δεν, πρόκειται να, δεν θα μπορέσει να προσέλθει στη συνάντηση αυτή, αλλά θα μας στείλει έναν βαθμό αξιωματούχο. Μην το πάρετε της μετρητής αυτό. Θα δούμε ποιος θα έρθει και βέβαια θα τον ε, βάλουμε με ερωτήσεις. Όσοι τώρα όσες γνωμοδοτήσεις έχουν γίνει για το έργο μας για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές δηλαδή όλες οι γνωμοδοτήσεις τις έχετε σίγουρα ένα αρκετά χοντρό βιβλίο και μεγαλώνει και άλλο τώρα μάλιστα την Παρασκευή που μας πέρασε λάβαμε επιστολή από την Επιτροπή Εξωτερικών και θα περιληφθεί και αυτή επομένω. Τελευταία δε ανακοίνωση στην συνάντηση της 1ης Φεβρουαρίου είχαμε έναν αριθμό συναδέλφων που δεν μπόρεσαν λόγω χρόνου, δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ερωτήσεις στον Επίτροπο, τις υπέβαλαν γραπτός. Η γραμματεία της Επιτροπής μας τις διαβίβασε αρμοδίως και σήμερα έχουμε τουλάχιστον τι απαντήσει του Επιτρόπου Έτιγκερ. Τις λάβαμε δηλαδή την Παρασκευή. Εγώ όμως σήμερα μόλις έλαβα γνώση. Τέλος πάντων είναι εδώ οι απαντήσει και όσοι είχαν υποβάλει ερωτήσει τις έχουν ήδη λάβει. Ας έρθουμε λοιπόν στο, τώρα στο ε, κυρίω θέμα της ε, ε διαταξίσμας που αναφέρεται στο σύστημα των ιδίων πόρων, όλοι και όλες, τουλάχιστον οι περισσότεροι, συμμετέχουμε ήδη από καιρού στα ευρωπαϊκά θέματα και ασχολούμαστε με το σύστημα ιδίων πόρων και από καιρό λέμε ότι απαιτείται μεταρρύθμισή του. Ειδικά σήμερα, μάλιστα, προς πληροφόρησή σας το λέω, διεξήγαγα συζήτηση περί ενός παραδοσιακού ιδίου πόρου, δηλαδή της εισφοράς ζαχάρεως και ισογλυκόζης. Δηλαδή χρειάστηκε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα και έμαθα ότι οι εισφορές αυτές κατά κάποιο τρόπο είναι δευμεσμένοι πόροι, είναι assigned revenues. Μέχρι το 6 σίγουρα, όπου ήταν και η μεταρρύθμιση της αγοράς και μέχρι το 8 που έγινε η μεταβατική περίοδος ήταν τα χρήματα που έρχονταν από την αγορά ζάχαρης, οι σφορέ αυτές δηλαδή που σπράττονταν από την αγορά ζάχαρης, πήγαιναν συγκεκριμένα για επιδοτήσεις εξαγωγών. Δηλαδή ξαναπήγαιναν στον, αγορά, στην, στον τομέα τη ζάχαρη. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Η αναδιάρθρωση του τομέα της αγοράς ζάχαρης, πληρώθηκε από τον ίδιο τον τομέα της ζάχαρης, το ταμείο έχει κλείσει πλέον αυτό, το 12 ούτως ή άλλως θα λήξουν όλα αυτά, θα υπάρχει και ένα πλεόνασμα το οποίο θα εισρεύσει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα είναι της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό είναι το ένα πράγμα, και βέβαια όλοι όσοι ασχολούνται με την ζάχαρη λένε δεν θέλουμε πλέον οι εισφορές μας να θεωρούνται ήδη πόροι. Ίσως και αυτό χρειάζεται να το συζητήσουμε, όταν δηλαδή θα συντάξουμε πια την έκθεσή μας. Οι ήδη πόροι δεν είναι και πολλοί, και ιδίως οι παραδοσιακοί. Γνωρίζετε ότι είναι και αναλόγως με την παραγόμενη ποσότητα ζάχαρης μέσα σε ένα χρόνο, αν έρχονται οι φόροι αυτοί στα 135 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, και εγώ σκέφτηκα ότι έχουν κάπου δίκιο, εφόσον έχει αλλάξει νομοθετικά η κατάσταση, πρέπει να δούμε εάν πραγματικά μπορούμε να εισπράττουμε τις φορές τους, αυτούς, τις φορές τους αυτές. Διότι, εκτός των άλλων, η εισαγόμενη ζάχαρη δεν πληρώνει τις φορές αυτές. Άρα, θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Τέλος πάντων, τώρα απευθύνω Πρωτίστως το καλώς ορίσατε στον Επίτροπό μας κύριο Λεβαντόφσκι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν είναι βεβαίως και η πρώτη φορά. Είναι ο άνθρωπός μας στην Κομισιόν κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι. Χαιρόμαστε που είναι πάλι εδώ κοντά μας. Πριν όμως λάβει τον λόγο ο Γιάννους Λεβαντόφσκι, τον λόγο θα βάλει ο Σαλβαδόρ Γαρίγα. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Λεβαντόφσκι, που σας γνωρίζουμε πολύ καλά και συνεργαστήκατε επί μακρόν σε αυτή την Επιτροπή. Γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης δαπανών και της πολιτικής δαπανών, στα πλαίσια του ΣΟΥΡ, δεν μπορούμε παρά να στραφούμε και στα έσοδα. Διαφορετικά θα προβαίναμε σε μία ανισόρροπη ανάλυση της δημοσιονομικής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Όπως είπε και η Πρόεδρος, από πλευράς πόρων βρισκόμαστε σε μία δυσχερή κατάσταση γιατί αφού αναλύσαμε τις δαπάνες θεωρήσαμε ότι για να διατηρήσουμε τις παρούσες πολιτικές, ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να μειωθεί. Επειδή υπάρχει βασική θέληση από ορισμένα κράτη-μέλη να μειώσουν την εισφορά τους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέλησή μας, τη θέληση του Κοινοβουλίου για μια αναθεώρηση των πόρων. Όπως είπε και η Πρόεδρος Χάουγκ, Μιλάμε για μια πολιτική κρίση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα υπολοιματικά ποσά και ως προς το ΦΥΠΙΑ, που είναι η τρίτη πρόσοδος, δεν τηρεί τα κριτήρια κοινής φορολογικής πολιτικής. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε νέα στοιχεία, όπως κάνει η Επιτροπή και ο κύριος Λεβαντόσκι μέσα στα πλαίσια του budget review που μας υπέβαλε εδώ και ορισμένους μήνες. Με την παρουσία του κυρίου Λεβαντόφσκι θα ήθελα να την εκμεταλλευτώ μάλλον για να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις αν και γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν πολύ πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αφού είδα την αντίδραση ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων, αρκετών εθνικών κοινοβουλίων, με τα οποία θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε κατά τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κοινοβούλια αυτά λένε ότι δεν θα πρέπει να μιλούμε για νέους πόρους, αλλά για αναδιάρθρωση των υπαρχόντων. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις εισφορές και την σχέση των εισφορών σε σχέση με το ΑΕΠ. Θεωρείτε, κύριε Λεβαντόφσκι, ότι μπορούμε να συμφιλειώσουμε και τις δύο θέσεις, δηλαδή να έχουμε έναν τέταρτο πόρο που είναι πιο διαφανής και να μην υπόκειται σε πολιτικές συζητήσεις κάθε φορά για καθαρές εισφορές ή καθαρούς εισφορείς. Ως προς το ΦΥΠΙΑ υπάρχουν ε, κοινοβούλια που ζητούν την εξαφάνισή του θα ήθελα να μας πει ο Επίτροπος κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί αυτό, αυτή η τρίτη πρόσοδος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες. Ως προς τους ίδιους πόρους, μέσα στα πλαίσια της εντολής ΣΟΥΡ, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα χρηματοδότησης που να βελτιώσει την δημοσιονομική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια ε, μιας μεγαλύτερης ορατότητας. Η Επιτροπή στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναθεώρησης μιλά για νέους σπόρους, ενδεχόμενους νέους σπόρους. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σε ορισμένους τομείς περισσότερο από ό,τι άλλους, άρα θα θέλουμε να ρωτήσουμε τον Επίτροπο ποιους ίδιους πόρους, ποιοι ίδιοι πόροι είναι οι πλέον κατάλληλοι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους νέους πόρους έτσι ώστε να είναι συμβατοί με την φορολογική αυτονομία και κυριαρχία των κρατών μελών. Επίσης, τι γνώμη έχει ο Επίτροπος ως προς τους ε, δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόστηκαν στις τρέχουσες ε, δημοσιονομικές προοπτικές μέσα στα πλαίσια του συσχετισμού ε, εισφοράς ωφελίας. Γιατί η ΣΟΥΡ μιλά για παλιφή μηχανισμών διόρθωσης, είτε πρόκειται για ταμεία ή πόρους ad hoc ή ε, πόρους μέσα στα πλαίσια ελεγκτικών μηχανισμών. Μέσα στα πλαίσια μιας τελικής πρότασης Επιτροπής ΣΟΥΡ. Ποτέ δεν μιλήσαμε για νέο ορισμό των ιδίων πόρων. Θεωρούμε ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει. Μιλάμε για ετήσιες όροφες σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Μιλάμε για 1,24% σε σχέση με το ΑΕΠ και νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα εντάξουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σε αυτούς τους άξονες θα μπορούσαμε να κινηθούμε και ελπίζουμε ο Επίτροπος να μπορέσει να μας αναπτύξει περισσότερο αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ίδιους πόρους που θα εντάξουμε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Σας ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Εσείς, Γιάννους, παρακαλώ, έχετε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να συζητώ μαζί σας, που δεν είναι η πρώτη βέβαια φορά, για το ευαίσθητο αυτό ζήτημα των ιδίων πόρων. Πρέπει να πω στα μέλη της Επιτροπής αυτής ότι όντως έχουν γίνει κάποιες πρώτες απόπειρες για την αναθεώρηση του συστήματος αυτού και ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη εντολή του και μάλιστα όταν ο κύριος Λαμασούρ είχε την πρωτοκαθεδρία τότε για την επανεξέταση του ζητήματος αυτού γίναν οι πρώτες προσπάθειες για να προλιανθεί το έδαφος αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε μια βαθύτερη μεταρρύθμιση. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις του Σαλβαδόρ Γκαρίγκα, θα μπορούσα να απαριθμίσω όλα τα δύνατα σημεία του υφισταμένου συστήματος, αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω αυτή τη στιγμή κάποιες εξηγήσεις, εφόσον όλοι γνωρίζετε για ποιο λόγο το σύστημα δεν είναι αρκετά διαφανές, για ποιο λόγο είναι πολύπλοκο και για ποιο λόγο δεν ευθυγραμμίζεται με τους πολιτικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται τελικά ότι ορισμένα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι οι δικέ τους δεν ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή όσον αφορά άλλα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά καταρχάς το ζήτημα της απλούστευσης. Πρέπει να σας πω ότι η απλούστευση αυτή θα πρέπει να περάσει από τα σημεία αυτά τα οποία έθιξε ο Σαλβαρό Γκαρίγκα. Ο ίδιος πόρος ο οποίος βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας δεν έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Είναι ένας αυθαίρετος ιδίο, ίδιος πόρος που βασίζεται απλώς σε κάποιες στατιστικές μελέτες. Επομένως η κατάργηση αυτού του πόρου πιστεύω ότι θα απλουστεύσει το όλο σύστημα των ιδίων πόρων και αυτή είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο εύκολο στο όλο εγχείρημα. Όσον αφορά τώρα τους νέους ίδιους πόρους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθότι υπάρχουν πολλές ευαισθησίες σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το ζήτημα της δημοσιονομικής κυριαρχίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν βάλουμε κατά της δημοσιονομικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Χρειάζεται μια ομόφωνη βάση συμφωνίας για οποιαδήποτε μελλοντική εισφορά στον κοινοτικό προπολογισμό και προφανώς και τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Μέλους θα πρέπει να εγκρίνουν μια νέα απόφαση στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναθεώρησης της, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρωθήκαμε σε έξι εναλλακτικέ λύσεις. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνανε πολλές ε, αναλύσεις, μελέτες τεχνικής φύσεως. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πάρα πολλά στοιχεία, τόσο πολιτικά όσο και τεχνικά, για τις έξι αυτές συναλλακτικές λύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στην ερώτηση του Σατβαδρό Γκαρίγκα και δεν μπορώ να πω τελικά ποιος έχει επιλεχθεί, ποιος νίκησε. Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό μόνο για αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες Μπορούμε πάντως σε κάθε περίπτωση να συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά των έξι αυτών υποψήφιων λύσεων. Ψάχνουμε το πιο αυτόνομο μηχανισμό, το πιο αυτόνομο εργαλείο, αυτό δηλαδή το οποίο δεν θα χρειαστεί να περάσει από τις εθνικές διοικήσεις για να συλλεχθεί. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό υποστήριξης του κοινωνικού προπολογισμού, ο οποίος θα είναι διασυνοριακός και αυτόνομος. Θα πρέπει να συνδέεται με το κοινοτικό κεκτημένο προς όφελος εσωτερικής αγοράς και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση οποιοδήποτε άλλου υποψήφιου ιδίου πόρου και πώς θα μπορούσε να ενισχύσει διάφορους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι ε, όλα αυτά ουσιαστικά επηρέασαν τις αποφάσεις που λάβαμε για την αθεώρηση των ιδίων πόρων την τελευταία εβδομάδα του ε, Ιουνίου. Αυτά έχω να πω αυτή τη στιγμή. Η Γιούτα ε, Χάουγκ μου έθεσε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό δεν μου επιτρέπει αυτό να δώσω πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες. Πάντως, όσον αφορά την επιλογή και την αξιολόγηση των υποψήφιων λύσεων, ε, το πιο σημαντικό να δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν από πολιτική πλευρά στη σημερινή Ευρώπη, η οποία πλήττεται από την κρίση, η οποία θα περάσει σε μια περίοδο πλέον μετά την κρίση και όσον αφορά το ζήτημα των διορθώσεων, ε, ζήτημα το οποίο έθιξε ο Σαλβαδόρ Γκαρίκα, ως προς αυτό έχω να πω το ακόλουθο. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών, ποιες είναι οι γυρικές τους δαπάνες, ποιες είναι οι δαπάνες όσον αφορά την συνοχή, ποιες είναι οι λοιπές δαπάνες των κρατών μελών. Θέλουμε να καλύψουμε δηλαδή όλο το τμήμα των δαπανών. Διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν αν δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τα ωφέλη των κρατών μελών. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε Πώ μπορεί να είναι πιο ισότιμο ο προπολογισμό και για τα 27 κράτη-μέλη σε όλου του τομεί του κοινοτικού προπολογισμού. Πρέπει επίση να δούμε πώ μπορεί να ευθυγραμμιστεί περισσότερο ο προπολογισμό και ο σχεδιασμό του με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είμαστε περισσότερο διαλλακτικοί, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ακούσουμε τις απόψεις όλων των συμβαλόμενων μερών, θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας συστάσεις και είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την μεταρρύθμιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η εκτίμηση μου αυτή είναι καθαρά ρεαλιστική. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δράσει μεμονωμένα. Υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία ε, έχουν ταχθεί υπέρ της μεταρρύθμισης του κοινοτικού προπολογισμού, αλλά η ουσιαστική μεταρρύθμιση και όχι μόνο η απλούστευση, η ουσιαστική μεταρρύθμιση θα περάσει από την δράση, την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά είχα να σας πω εισαγωγικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα σχόλιο μόνο θα ήθελα να κάνω. Πρωτού ακούσουμε και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα ευθύ αμέσως να πω το εξής. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην παραδοσιακή αυτή συζήτηση για τους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς αποδέκτες. το ζήτημα αυτό ουσιαστικά βάλει κατά τη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν μα συμφέρει να μιλάμε για το ζήτημα αυτό. Δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α εγκαταλείψουμε επιτέλου αυτή την οπτική γωνία, η οποία είναι καθαρά αρνητική. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα προ το Συμβούλιο και στους εκπροσώπους του που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, θέλουμε επιτέλους να σταματήσουμε αυτή την καταθλιπτική συζήτηση για τους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς αποδέκτες. Το ΕΛΚ πρώτο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα εισαγωγικά του λόγια. Όπως είπε και ο Επίτροπος, Από τη μια, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε το τρέχον σύστημα, θα πρέπει να του δώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και όπως είπε, η όλη συζήτηση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύκολη, αλλά αν πραγματικά θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτε να πλησιάσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταλάβουν καλύτερα πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη απλούστευση και μεγαλύτερη διαφάνεια στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε έναν καλό προπολογισμό που θα γίνεται κατανοητό από του πολίτε και θα είναι ένα προπολογισμό με μεγαλύτερα έσοδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ετήσιο προπολογισμό, αλλά θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει ένα κείμενο στο οποίο θα φαίνεται ξεκάθαρα από πού έρχονται τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε σε θέση να έχουμε το κείμενο αυτό, να το συζητήσουμε στη συνέχεια και θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των συζητήσεων που θα γίνουν επί του προπολογισμού. Ο Επίτροπο αναφέρθηκε σε μια σειρά πλουστεύσεων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα, για παράδειγμα κατάργηση του ίδιου πόρου που βασίζεται στο φόρο προσθέμενης, στο φόρο προσθέμενης αξίας, το μέτρο αυτό να προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια στον κοινοτικό προπολογισμό και δεχομένω να καταφέρουμε να ξεκαθαρίσουμε και λίγο την κατάσταση με τι πολλέ διορθώσει και επιστροφέ προβλέπονται για ορισμένε χώρε. Όσον αφορά τώρα τον, την κατάργηση του ιδίου πόρου που βασίζεται στο φόρο προστιθέμενη αξία. Ω προ αυτό πιστεύω ότι θα δοθεί σαφώ μια μεγαλύτερη διαφάνεια στον κοινοτικό προπολογισμό και σύν της άλλη, θα ξεκαθαριστεί όλη η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για το φόρο προσθέμενης αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε τις βασικές αρχές της συνθήκης της Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λέγεται ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτείται από ιδίους πόρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, μια σημαντική συμβολή στον κοινοτικό προπολογισμό η οποία γίνεται μέσω ιδίων πόρων και η οποία στη συνέχεια επιστρέφεται μέσω του συστήματος διόρθωσης και επιστροφών, δεν είναι κάτι το θετικό. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο, κυρία Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση της συζήτησης είναι να σταματήσουμε την αένεια αυτή συζήτηση που γίνεται για καθαρούς εισφορείς και καθαρούς αποδέκτες Αν κατάλαβα καλά στη συνέχεια τόσο είπε ο Επίτροπος, Μα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μακροπρόθεσμες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση των πολιτικών αυτών. Νομίζω ότι όντω αυτό είναι ο καλύτερο. Ε, το, η καλύτερη δυνατή λύση την οποία θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε πλέον στον ίδιο πόρο που βασίζεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Βέβαια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε να δημιουργηθεί εντύπωση στον νέο κοινοτικό προπολογισμό ότι δημιουργούμε νέους φόρους σε κοινοτικό επίπεδο και ας βασιστούμε περισσότερο στα όσα έχει πει ο κύριος Λαμασούρ στη δική του έκθεση που έθεσε τις διαφορετικές συνιστώσεις του νέου αυτού φόρου. Ένας φόρος ο οποίος θα πρέπει να είναι καθαρά ουδέτερος. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σημαντικότερος στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχουμε. Θα πρέπει επίσης να μειωθούν κατά κάποιον τρόπο και με ένα ξεκάθαρο τρόπο οι εισφορές των κρατών μελών. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας αυτό το περίφημο «juste είναι πια ξεπερασμένο. Δεν θα πρέπει να δεχθούμε ποτέ κάτι τέτοιο. Σεις έχετε το λόγο. Κύριε Λεβαντόφσκι, εδώ βρίσκεστε για, μια άλλη φορά, για άλλη μια φορά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν περίμενα να μου πείτε ποιος θα κερδίσει αυτά τα δημοσιονομικά έπαθλα αλλά ήθελα να μας δώσετε ορισμένες λεπτομέρειες σε σχέση με τους έξι υποψηφίους για ένα καλύτερο δημοσιονομικό μέσο. Αυτοί οι έξι υποψήφοι είναι αυτοί που εμφανίστηκαν στο budget review εδώ και μερικούς μήνες και τότε σας είχαμε υποβάλει το ερώτημα γιατί σας είπαμε ότι αυτός ο φόρος ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι πολύ σημαντικός για τους σοσιαλιστές. Μας είπατε ότι δεν θα τον απαλείψετε αυτό το φόρο, ότι υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές υπό εξέταση, αλλά ανάμεσα στους έξι υποψηφίους θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Ποιοι είναι αυτοί ότι οι έξι υποψήφοι για το Όσκαρ του καλύτερου δημοσιονομικού μέσου. Και επί ποιων στοιχείων εργαστήκατε για να θέσετε πιτάπιτος ορισμένους και να απομακρύνετε άλλους. Γιατί από το budget review φαινόταν ότι η Επιτροπή είχε κάποια προτίμηση για τους ε, ε, για τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ίδρυμα σε σχέση, ιδρύματα σε σχέση με αυτό τον φόρο χρηματοπιστών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και δεν κατανοούμε και θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του μεν ή του δε. Δηλαδή, οι φόροι αυτοί είναι εντελώς διαφορετικοί και αυτό αφορά όλους τους τύπους φόρων. Είτε πρόκειται για τον άνθρακα, είτε πρόκειται για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή φόρους ακινήτων. Όλα έχουν, όλοι έχουν τα υπέρ και τα κατά. Μερικοί θα μπορούσαν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Έτσι ώστε να ε, φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτό το θέμα των ε, ίδιων πόρων. Μιλήσατε για προαπαιτούμενα για, αυτούς τους, ε, για αυτό το μηχανισμό. Καταρχήν, αυτοί οι δημοσιονομικοί μηχανισμοί θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί. Δεν θα πρέπει κανείς να κάνει ε, δημιουργικές λογιστικές ή να προβάλλει ταχυδακτηλουργικούς ε, μηχανισμούς ή ελιγμούς και εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να καταβάλουν αυτή την εισφορά οι πολίτες. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία γιατί ισχύει ο μεν και όχι η δε. Σας ευχαριστούμε. Όντως έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το, το χρονόμετρο ο τεχνικό πίσω μα δεν επιτρέπεται ούτε να αγγίξει το χρονόμετρο. Δεν το σχολιάζω αυτό. Άλλη υπηρεσία είναι αρμόδια και αυτή η υπηρεσία δεν τα έχει κάνει σωστά. Αλλά έχει το handy τη εδώ η Μόνικα, έχει δηλαδή το κινητό τη τηλέφωνο, το οποίο έχει και κάποιο είδο ε, χρονόμετρο, μάλιστα και με δευτερόλεπτα. Άρα ε, μετρά το χρόνο και έντα τα πήγε πολύ καλά. Χάγκλουντ, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ ωραία, τα, ε, ωραία χρονομετρείτε τον χρόνο της ομιλίας μας πολύ γερμανικά. Ευχαριστώ πρώτα τον Επιτρόπο που είναι παρόν. Στην πολιτική μας ομάδα μας ικανοποιεί η συζήτηση αυτή και βλέπουμε θετικά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά δηλαδή στη, με τη συζήτηση για τους ιδίους πόρους. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις που θα υποβάλλετε την Άνοιξη και το καλοκαίρι. Κατανοώ ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις του κυρίου Γκαρίγα. Εγώ θα σας υποβάλω όμως μερικές ακόμη προς την ίδια κατεύθυνση, να δω ποιες θα μπορέσετε να απαντήσετε. Η αντικατάσταση πρώτα της ε, φορολογικής βάσης του ΦΠΑ σχεδιάζεται να ε, υποβάλλετε προτάσεις για νέους ιδίους πόρους που θα είναι συμπληρωματικοί ε, επιπλέον του ΑΕΠ ή θα προτείνετε νέους ε, πόρους που θα αντικαταστήσουν την, ε, την εισφορά στη βάση του ΦΠΑ. Αν απαντήσετε θα είναι χρήσιμο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε προς τα πού κατευθύνεται η σκέψη σας και ποιο είναι το μέρος του προϋπολογισμού που νομίζετε ότι μπορεί να καλυφθεί με τους νέους αυτούς πόρους, ίσως και το 100% θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Σε ό,τι, αφορά τώρα ουδέτερους ίδιους πόρους, είναι νομίζω αφελές να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να, είναι, να υπάρχει ουδέτερος ίδιος πόρος. Λέμε να μην φορολογήσουμε τους πολίτες. Ας μην λησμονούμε ότι σε βάθος χρόνου όλα επηρεάζουν τους πολίτες. Για παράδειγμα, εάν φορολογηθούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, έμεσα θα επιβαρυνθούν εν τέλει οι πολίτες, γιατί θα κρυβίνουν οι συναλλαγές αυτές για τους πολίτες. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να το έχουμε πάντοτε η υπόψη μας. Σχετικά με ορισμένους ιδίους πόρους είναι πολύ επιφυλακτική η πολιτική μας ομάδα σε ό,τι αφορά την μνήα ορισμένων ιδίων πόρων. Πάντως συμφωνούμε με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την διενέργεια μελέτης επιπτώσεων πρώτα. Εάν μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο τι μπορείτε να προτείνετε σε ό,τι αφορά τέλο πάντων το χρήμα. Και θα ήταν χρήσιμο εν τέλει να σχολιάσετε και το επίπεδο θάρρους που μπορεί, στο οποίο μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είδαμε τελευταία μία τάση που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά θαραλέα και φοβούμαστε κι εμείς ότι εάν αντιμετωπίσετε πολλή αντίσταση από το Συμβούλιο δεν θα έχετε το θάρρος, δεν θα έχετε τα κότσια να σπρώξετε αρκετά τις ε, προτάσεις αυτές. Θα μπορούμε λοιπόν να αναμένουμε θαραλείς προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστω και αν υπάρχει αντίσταση από το Συμβούλιο. Γιούτα Χάουκ. Ναι, αλλά ελπίζω ότι όλοι ενθαρρύνουμε τον Επίτροπο στην πορεία του αυτή. Ιζαμπέλ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλη η συζήτηση για τους ιδίους πόρους αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την κοινοτική αυτή νομοθεσία για τον κοινοτικό προπολογισμό τόσο για μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εντοπιστούν οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι σε σχέση με αυτά που είπατε και σε σχέση με αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου πριν από μένα. Να πω καταρχάς ότι το ζήτημα των καθαρών εισφορών και των καθαρών αποδεκτών είναι μια συζήτηση που δεν μας αρέσει, που ουσιαστικά δεν συνάδει καθόλου με τα όσα επιθύμησαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση αυτή. Όσον αφορά τους καθαρούς εισφορείς, θα πρέπει να προσέξουμε να μην ξεκινήσουμε πάλι μια συζήτηση για τις δαπάνες, για τα περιθώρια, όπως είχαμε κάνει το 2005, όπου ουσιαστικά έγινε μια προσέγγιση μόνο σε εθνικό επίπεδο και προσπάθησε κράτος, κάθε κράτος μέλος να δει πώς θα καταφέρει να προσαρμόσει καλύτερα για το δικό του συμφέρον τον κοινοτικό προπολογισμό. Δεν θα ήθελα να μας ανακοινώσετε ποιοι νίκησαν στα Όσκαρ, κύριε Επίτροπε, γιατί πριν τους νικητές είχαμε τους υποψήφιους. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υποψήφοι. Πριν από λίγο αναφερθήκατε απλώς σε κάποια κριτήρια. Κάνατε μια κάποια ανάλυση, είπατε το διασυνοριακό αναφερθήκατε στον διασυνοριακό χαρακτήρα, είπατε ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν οι εθνικές διοικήσεις, είπατε ότι θα πρέπει τα νέα αυτά μέτρα να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο. Μάλλον δεν μπορείτε να μας πείτε πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα. Θα πρέπει πάντως να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοί σα. Και χρειαζόμαστε και εμείς πληροφορίες από εσάς για την εργασία την οποία κάνετε. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να έχετε τη δική μας υποστήριξη. Την υποστήριξη του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ιδίω σε σχέση με το Συμβούλιο, όπου είδαμε ότι ε, ο όρος ε, ήδη πόρη στο Συμβούλιο προκαλεί πάρα πολλές φορές πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τι κάνετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε. Χρειάζεστε και εσείς εμάς και εμείς σας χρειαζόμαστε. Εξαρτώμεθα λοιπόν από εσά για να μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες και για να εργαστείτε μαζί, μαζί Επίσης, θα ήθελα και εγώ να πω ότι θα πρέπει όντως να υπάρχει αυτό το επίπεδο ουδετερότητας στον κοινοτικό προπολογισμό. Δηλαδή, οτιδήποτε αποφασίσουμε θα πρέπει να οδηγεί σε μικρότερες δαπάνες για τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και ξέρετε πώς έχουν οι εθνικοί προπολογισμοί αυτή τη στιγμή. Οι περισσότερες χώρες περνάνε από πάρα πολύ δύσκολες περιόδους. Το Μάρτιο το Συμβούλιο θα συζητήσει για μια οικονομική κατάσταση που δεν είναι καθόλου εύκολη για κανένα κράτος μέλος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο θα συνάδει με τα μέτρα τα οποία περιγράψετε εσείς και θέλουμε και ε, ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα είναι ευνοϊκά για τα κράτη-μέλη. Κατά αυτόν τον τρόπο και η δική σας εργασία θα είναι πιο εύκολη και θα Επιτρέψτε κατά αυτόν τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργεί την περίφημη αυτή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι δική μας την βούληση καταρχάς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταφέρουμε να συνεργαστούμε το συντομότερο δυνατό για τα σημαντικότητα αυτά ζητήματα των ιδίων πόρων. Άλλωστε, στα πλαίσια του ε, προϋπολογισμού του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούμε ακριβώς να δούμε πώς θα καταφέρουμε να δαπανίσουμε λιγότερα χρήματα για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να πετύχουμε και εμείς ένα κάποιο επίπεδο προστιθέμενης αξίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τόσα μας είπατε και για τόσα θα μας πείτε κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ισαβέλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και σε αυτό οφείλει να εγκύψει ο Επίτροπος. Ο κόσμος έξω δεν καταλαβαίνει πώς εισπράττονται τα χρήματα και από τη δική μου οπτική γωνιά το γεγονός ότι έχετε ένα σύστημα επιστροφών δείχνει ότι υπάρχει κάπου ε, μια έλλειψη δικαιοσύνη στο σύστημα. Εγώ δέχομαι ότι αυτό χρειάζεται διόρθωση και δέχομαι να υποβληθούν ιδέες. Τώρα πρέπει να δούμε σε τι συμφωνούμε. Να αλλάξουμε, να αντικαταστήσουμε τον ένα μηχανισμό ιδίων πόρων με έναν άλλο, δεν νομίζω να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Και δεύτερο, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομική ανεξαρτησία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος και της ενιαίας αγοράς και της κοινής αγροτική πολιτικής. Γι' αυτό το υποστηρίζουμε το σύστημα αυτό. Από την άλλη μεριά έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις με τη συνιστόσα που προέρχεται από τον ΦΠΑ. Εδώ υπάρχει έλλειψη διαφάνεια και ασφαλώ χρειάζεται μεταρρύθμιση. Δεν είμαι ωστόσο πεπισμένο σχετικά με του άλλου υποψηφίου, Δύο εν προκειμένου, φόρος επί των, δημοσιονομικών επί των ε, οικονομικών συναλλαγών και ο φόρο επί των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Ήδη η χώρα μου έχει σημαντική, σημαντικό πρόβλημα και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο με τα συνδικάτα, εάν συνεχίσουμε προ την κατεύθυνση αυτή για το διορθωτικό μηχανισμό. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να βγάλουμε από τη μέση τα συναισθηματικά σχετικά με τις επιστροφές και δούμε τα μαθηματικά, διότι πρόκειται περί απλών μαθηματικών. Στο κάτω της γραφής είναι απόδοση δικαιοσύνης και η θετική πλευρά είναι ότι ταυτόχρονα είναι και μια, ένα κίνητρο για τις χώρες μέλη να μην εξαντλούν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και τέλος για ε, το στοιχείο που βασίζεται στο ΑΕΠ, τη συνιστόσα δηλαδή που βασίζεται στο ΑΕΠ. Η Ένωση είναι αυτή η οποία εξαρτάται από τις χώρες μέλη. Αυτό είναι ο χαρακτήρας. Βάζοντας τη συνιστόσα αυτή του ΑΕΠ, επιτρέπει, επιτρέπεται έτσι στις χώρες μέλη να διατηρούν τον έλεγχο για το μεγαλύτερο μέρος του κοινωτικού προϋπολογισμού και επομένως μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστούμε. Μιγγέλ Πόρτας. Ευχαριστώ. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ο Επίτροπος έρχεται για να συζητήσουμε τα θέματα περί πόρων χωρίς να έχει κανένα νέο επιχείρημα, πρόταση ή νέα ιδέα ούτε καν αξιολόγηση των προγενέστερων προτάσεων. Άρα είναι μη παραγωγική αυτή η συζήτηση. Βεβαίως ο Επίτροπος κατέχει την τέχνη του να μην απαντά, αλλά εδώ θα πρέπει, θα πρέπει να συζητήσουμε για ε, Όσκαρ ρητορίας εδώ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μας μίλησε για 10 λεπτά και δεν μάθαμε τίποτα το καινούριο. Μπορώ να πω κι εγώ ορισμένα πράγματα από τη δική μου πλευρά. Το παρόν σύστημα είναι παράλογο. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου τα κράτη θέλουν να εισφέρουν με το λιγότερο και να λαμβάνουν το περισσότερο δυνατόν. Άρα δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του αυτός ο μηχανισμός, άρα θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμφωνούμε επ' αυτού. Επίσης, οι ίδιοι πόροι δεν μπορούν να επικεντρώνονται στο ΦΠΑ, γιατί τότε δεν είναι ήδη πόροι. Άρα, υπό το φως των εργασιών του ελεγκτικού συνεδρίου, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή μέσω ΦΠΑ που όπως κρίνει το ελεγκτικό βρίσκεται στην τάξη των 200 δις ευρώ. Δηλαδή το διπλό του παρόντος προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να συζητάμε για το ΦΠΑ αν θα μιλήσουμε για την φοροδιαφυγή καταρχήν. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι άκουσα πολλές επικρίσεις για έναν φόρο για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά το μόνο επιχείρημα που άκουσα είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μετακύλιαν αυτή την εισφορά στους ε, πελάτες, στους καταναλωτές. Άρα Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τα ασφαλιστικά ιδρύματα, διότι μετακυλίεται αυτό το κόστος πάντα στον πελάτη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μετατρέψουμε τους πόρους σε έναν ε, ε, μοχλό κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακατανομής που να οδηγήσει σε μια κοινωνική δικαιοσύνη. Θα πω στον Επίτροπο το εξή. Το Κοινοβούλιο έλαβε μια θέση κατά των φορολογικών παραδείσων. Μιλήσαμε, μάλλον καταδικάσαμε τους φορολογικούς παραδείσους. Ολοκληρωτικά. Πότε θα εντάξετε τους φορολογικούς παραδείσους επίσης στο μηχανισμό των Όσκαρ που μας προτείνατε. Ακολουθεί η κυρία Τζαβέλα. Α, α, όχι, όχι. Η κυρία Αντριάσιν. Νομίζω ότι η όλη συζήτηση για τους ιδίους πόρους είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή, εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουμε από τους πολίτες να συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστες πληροφορίες. Δεν ήμουν εδώ από την αρχή της συνεδριασής μας. Πάντως δεν πιστεύω ότι ο Επίτροπος Λεβαντόσκι κατάφερε να αποσαφηνίσει κάποια σημαντικά στοιχεία της όλης συζήτησης. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε σε έξι υποψηφίους όσον αφορά τους νέους ίδιους πόρους. Ξέρω ότι μιλήσατε για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το φόρο επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι όμως υποψήφοι για τους ίδιου πόρους. Επίσης, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Κάνετε κάποια μελέτη αντικτύπου για, τον κάθε έναν, για την κάθε μία από τι εναλλακτικέ αυτέ λύσει, όσον αφορά δηλαδή τον καταναλωτή, όσον αφορά τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και αν κάνετε μία τέτοια μελέτη, θα μα δώσετε τότε και τα αποτελέσματα και τα αριθμητικά στοιχεία, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμεί τη δική μα αξιολόγηση αντικτύπου. Τρίτη ερώτηση. ποιες είναι οι διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις που μπορούν να υπάρχουν σε σχέση με κάποιους φόρους. Θα ε, περιμένετε από τα κράτη-μέλη πάλι να έρθουν κάποιες εισφορές ή θα πρέπει αυτές οι νέες εισφορές να γίνουν πλέον από τις Βρυξέλλες σε κοινοτικό επίπεδο. Και ποιες ήταν οι διαπραγματεύσεις ω προ τον προπολογισμό, αν είμαστε σε θέση εμεί άμεσα να συγκεντρώνουμε του ε, ίδιου πόρου και ποιο θα είναι υπεύθυνο για την απαλλαγή στην περίπτωση αυτή, αν καταφέρουμε άμεσα να συγκεντρώνουμε ίδιου πόρου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο Χάουκ. Πριν δώσω τον λόγο πάλι στον Γιάννου Λεβαντόφσκι για να απαντήσει ξανά, να πω μόνο το εξή σχόλιο. Αντί να του ριχνόμαστε του Επιτρόπου, καλύτερα να τον ενθαρρύνουμε. Δεν βρίσκω ότι είναι αλήθεια ότι μίλησε 10 λεπτά και δεν είπε τίποτα. Και το δεύτερο, όποιος ξέρει να διαβάζει, νομίζω έχει ένα πλεονέκτημα. Αυτό δηλαδή, με λίγα λόγια θέλω να πω ότι όλοι έχετε το budget review σε όλες τις γλώσσες. Και τους περιλαμβάνει εκεί τους έξι υποψηφίους ξεκάθαρα ορισμένου. Δεν θέλω βέβαια να μαλώσω του συναδέλφου μου, αλλά ασφαλώς χρειάζεται επίκριση και ο ίδιος ο Επίτροπος όταν αυτό, αυτή η επίκριση είναι δικαιολογημένη, αλλά εν προκειμένου νομίζω ότι δεν είναι. Γιάννους, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Γιούτα για την υποστήριξη. Ε, σας ευχαριστώ για τις ευφυείς αυτές ερωτήσεις σας. Και λέω ευφυείς γιατί προσπαθείτε αυτή τη στιγμή όντω να αποσπάσετε από μένα περισσότερε πληροφορίε από αυτέ που μπορώ εγώ να σα αποκαλύψω. Και ο κύριο ε, Πόρτα, μάλιστα, ε, με έναν βάναυσο τρόπο ουσιαστικά περιέγραψε το δεκάλεπ, τη δεκάλεπτη αρχική μου ομιλία. Συμφωνώ με τον Ζων ε, Λουκ και με την πολιτική ανάλυση ε, που έκανε του όλου αυτού περιβάλλοντος ε, τρεις ε, μήνες προτού ανακοινώσουμε ουσιαστικά τον νικητή, τον επιλεγμένο αυτόν ιδιωτικό, ε, ίδιο πόρο, που θα πρέπει αυτό να γίνει στα πλαίσια όλων αυτών των πολιτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, το στοιχείο της ουδετερότητας είναι, αν θέλετε, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην όλη πρόταση. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτεύουσες που θέλουν να μειωθεί η εθνική, η εθνική εισφορά. Αυτό όμως θα γινόταν αν ήμασταν πραγματικά σοβαροί όσον αφορά το ζήτημα της ε, ουδετερότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσαμε να μειώσουμε όμως τις, ε, τα άλλα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επηρεάζει ουσιαστικά και την αξιολόγηση του ίδιου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το να μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε έναν πραγματικό φόρο προστιθέμενης αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσε να τροφοδοτούσε και να ενίσχυε άμεσα τον κοινοτικό προπολογισμό. Είναι δύσκολο λοιπόν το ζήτημα της ουδετερότητας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε γνήσιους νέους ίδιους πόρους. Είναι δύσκολο σίγουρα αυτό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε την όλη αυτή προσπάθεια. Και Πιστεύω ότι όλες οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα πρέπει ουσιαστικά να σέβονται το πνεύμα των ευρωπαϊκών συνθήκων και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν εναντίον τους, όπως πολλές φορές γίνεται με την όλη συζήτηση για τους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς αποδέκτες. Ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών αναφέρθηκε σε έναν ίδιο πόρο, ο οποίος πιστεύω ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, που έχει να κάνει με τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχει αναλυθεί πάρα πολύ η εναλλακτική αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, θα μπορούσαμε να είχαμε έναν ίδιο πόρο που θα βασίζεται σε αυτές τις συναλλαγές και που θα μπορούσε να έχει μία ευρεία βάση, θα μπορούσε να καλύπτει διάφορες πολλές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή θα μπορούσε να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μόνο χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι και στα πλαίσια μία και μόνο αναλεκτικής λύση, δηλαδή για παράδειγμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, υπάρχουν πολλέ επιμέρου στη συνέχεια εναλλακτικέ που απαιτούν περισσότερες ακόμα αναλύσεις και μελέτες προκειμένου να δούμε τελικά τι μπορεί να γίνει στην πράξη και τι δεν μπορεί να γίνει. Και πέρα από τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αναφερθήκαμε και στο ζήτημα του φόρου των ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά εδώ πέρα αναφερόμαστε στις ε, μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες οι οποίες μετέχουν ενεργά στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πάντω, ο φόρος αυτός χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι μη εναλλακτική, αλλά ένας σημαντικός, αν θέλετε, νέος υποψήφιος ίδιο πόρο. Αναφερθήκαμε επίσης και στις επιπτώσει επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι υποψήφοι σε εθνικό, αλλά πολλές φορές και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν ε, επίσης να επηρεάσουν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητα σε κάθε χώρα και αυτό το ζήτημα το αναλύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον κύριο Χάκλουν και στις παρατηρήσεις του μία σύντομη απάντηση, εύκολη απάντηση θα ήθελα να δώσω. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουμε τόσο εύκολα την εθνική εισφορά που αντιστοιχεί στο 76% του προπολογισμού. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον το 1 τρίτο του προπολογισμού και βλέπω ότι συμφωνεί και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί δεν θα ήθελα να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και με τα οποία δεν θα συμφωνούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, η φιλοδοξία μας είναι τουλάχιστον το 1 τρίτο του προπολογισμού να μπορεί να χρηματοδοτηθεί διαφορετικά. Από την δεκαετία του 80 αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι οι εθνικές εισφορές δημιουργούσαν ένα είδος ισορροπία στον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά δεν καταφέρναμε ουσιαστικά να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στους ίδιους πόρους και τις εθνικές εισφορές. Οι εθνικές εισφορές, αν μη τι άλλο, καταφέραν να δώσουν μια σταθερότητα στον προπολογισμό και μας επέτρεπε αυτό να κάνουμε κάποιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Έπειτα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κουράγιο, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κότσια, όπως είπατε. Κοιτάξτε, Νομίζω ότι το δικό μας το θάρρος εξαρτάται από το δικό σας το θάρρος, από τα κότσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τη δική σας ουσιαστικά την αποφασιστικότητα να προχωρήσετε με νέα μέτρα για το μέλλον, για τον κοινοτικό προπολογισμό και όχι μόνο για τον, Ευρω... για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπάρχουν και διάφορα think tanks στις Βρυξέλλες, διάφορα κέντρα ανάλυσης που έχουν ήδη καταλήξει στο ότι θα προτιμούσαν να υπάρχει ένας κοινοτικό φόρος προστιθέμενης αξίας. Όλα αυτά τα think tanks όμως είναι απλώς κέντρα μελετών και ανάλυσης. Δεν έχουν κάποια πολιτική υπόσταση. Δεν μπορούν να δώσουν πολιτική πυγμή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια συνεννόηση, μια συμφωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουμε περισσότερο. Κυρία Ντιογόν τώρα αναφερθήκατε στα πράγματα που είπε και η Γιούτα στην αρχή. Είπατε ότι σε καμία περίπτωση θα πρέπει να επαναληφθεί όλη η συζήτηση που γίνεται από το Συμβούλιο για τους καθαρούς εισφορείς. Εμείς μιλάμε όμως αυτή τη στιγμή και για τις δαπάνες και χρειαζόμαστε τη δέσμευση και των 27 κρατών μελών. Και θα πρέπει επίσης να δούμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπο, ο ποσοτικό που θα έχουν οι νέε αυτέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 27 κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε εκτός της συζήτηση τη στάση των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε εντελώ τις εθνικές ανησυχίες. Ο κύριος Άσφορτ έχει δίκιο επίσης τα όσα είπε στη συνέχεια. Δεν μπορούμε εύκολα να αντικαταστήσουμε τον έναν ίδιο πόρο με κάποιον άλλον. Δεν είναι εύκολη η άμεση αντικατάσταση. Η Γιούτα αναφέρθηκε για παράδειγμα στην εισφορά ζάχαρης και ισογλυκόζης, μια εισφορά η οποία δεν συμβάλλει πάρα πολύ στον κοινοτικό προπολογισμό, αντιστοιχεί σε ένα μηδαμινό ποσοστό του κοινοτικού προπολογισμού. Από την άλλη όμως έχουμε τους τελωνιακούς δασμούς που αντιστοιχούν σε ένα 12% και οι τελωνιακοί αυτοί δασμοί θα επηρεαστούν και θα μειωθούν στο μέλλον κάθε φορά προχωράμε όλο και περισσότερο με την απελευθέρωση της αγοράς. Μια απελευθέρωση της αγοράς θα οδηγήσει σε μείωση των ελληνικών δασμών και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης του κοινοτικού προπολογισμού από τους ελληνικούς δασμούς. Όσον αφορά τώρα τα όσα είπε ο κύριο Πόρταν με αρκετά βάναυσο και βίαιο τρόπο για το πόσο απογοητευμένο ήταν από την αρχική δεκάλεπτη εισήγησή μου. Αυτή είναι όμως η τοποθέτησή μου σήμερα. Τι άλλο μπορώ να σας πω πέρα από αυτό. Επίσης αναφερθήκατε κύριε Πόρτα σε κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το όλο εγχείρημα δεν έχει να κάνει μόνο με την έβρεση νέων ίδιων πόρων, έχει να κάνει και με την ίδια την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή έχει... συνδέεται ήδη με τη συζήτηση που γίνεται για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θα καταφέρουμε να τυποποιήσουμε ακόμα και το φορολογικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μειώσουμε τα επίπεδα απάτης και φοροδιαφυγής. Δεν μπορώ και γι' αυτό να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Πάντως πιστεύω ότι ε, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας μπορεί να οδηγήσει και αυτό με τη σειρά του στη μείωση τη απάτη και στην αύξηση τελικά των ε, ιδίων πόρων. Επίση, αναφερθήκατε σε με ρωτήσατε ποιοι είναι οι έξι υποψήφοι διπόροι. πόροι. Είπαμε φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόρο επί των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, τέλο αεροπορικών μεταφορών, κοινοτικό φόρο προσθέμενη αξία, ένα συνεργειακό φόρο και ένα φόρο εισοδήματο εταιριών. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να έχουμε ένα διασυνοριακό χαρακτήρα σε αυτά τα τέλη και σε αυτούς τους φόρους. Ο διασυνορικός αυτός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το τέλος αεροπορικών μεταφορών. Ο κύριος Σόιμπλε έχει αναφερθεί στο ζήτημα αυτό και είχε πει ότι υπάρχουν ορισμένες γερμανικές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες είχαν συνειδητοποιήσει ότι είχαν ένα φορολογικό κίνητρο για να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να καταφέρουμε να θεσπίσουμε ένα τέλος αεροπορικών μεταφορών, το οποίο θα μπορεί να τροφοδοτεί με πόρους τον κοινοτικό προπολογισμό, ο οποίος όμως θα είναι δίκαιος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα οδηγεί σε αυθαίρετη μετατόπιση της έδρας των αεροπορικών εταιριών. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην μου κάνει νέα επίθεση ο κύριος Πόρτας. Ειλικρινά δεν, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ.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 τρία λεπτά ο καθένας και όχι τέσσερα. Πολλά θέματα έχουν καλυφθεί, Πρόεδρε, γι' αυτό θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Δύο πράγματα μου έκαναν, με εξέπληξαν ως προς τον προϋπολογισμό. Τη στιγμή που το 70% προέρχεται από την εισφορά των κρατών μελών, θα έχουμε μία μεγάλη μάχη κάθε χρόνο και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει ο επιμερισμός των ιδίων πόρων και ίσως αυτό επιλύσει εν μέρη το θέμα. Εάν δούμε το νέο σύστημα, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα νέο φόρο επί των ιδιωτών, δεν θα το δεχτούν αυτό και θα πρέπει να υπάρχει η δημοσιονομική ουδετερότητα ως προς την εισφορά των κρατών μέλων και οι περισσότεροι συμφωνούν επ' αυτού. Η μεγαλύτερη δυσκολία προέρχεται από το Συμβούλιο, από ορισμένα κράτη-μέλη, αν και δεν αρνούμε το θάρρος της Επιτροπής και φαντάζομαι ότι θα μας προβάλλει μια συγκεκριμένη εναλλακτική στο μέλλον. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον Επίτροπο κατά πόσο έχουν γίνει άτυπες ή μη συζητήσεις με τα κράτη-μέλη επί του θέματος, γιατί η Επιτροπή ΣΥΡ και η Επιτροπή θα πρέπει να επινοήσουν ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων με βάση μία ε, προτινόμενη εναλλακτική, την οποία και θα προτιμήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να μάθει από το Συμβούλιο τι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Διαφορετικά θα καταναλώσουμε πολύ φαιά ουσία και χρόνο και στο τέλος δεν θα φτάσουμε πουθενά. Σας ευχαριστώ κύριος Έλλης. Ορισμένες φορές καταλήγει κανείς να μην καταλαβαίνει. Στο δεύτερο παράρτημα του εγγράφου που μας δώσατε βρίσκω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί βλέπετε ότι ο πόρος του ΑΕΠ ήταν 1,2% το 1992 και το ίδιο μειώθηκε μάλλον τώρα, είναι γύρω στο 1. Νομίζω ότι αυτό ε, πρέπει να ενδιαφέρει τις χώρες μέλη. Ωστόσο, δύο ερωτήσεις, ε, κύριε Επίτροπε. Πρώτο, γιατί μετά την απόφαση του 1988 είδαμε σημαντική πτώση της συνιστώσεως του ΦΠΑ όπως λέει και το έγγραφό σας, είναι στο 11% του προϋπολογισμού το 2009. Γιατί μειώθηκε και ποιο είναι το πρόβλημα και ποιος θα ήταν καλός πόρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, η φράση που χρησιμοποίησατε για τις διορθώσεις. Στα αγγλικά το είπατε και άρα νομίζω ότι σωστά το, κατάλαβε, το κατάλαβα. Είπατε ότι πρέπει να παραμείνει εάν δεν λειτουργήσουν οι άλλες ε, λύσεις για, τα, για τις δαπάνες. Πώς θα πείσω εγώ τους ψηφοφόρους μου στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 2003 τους είχαμε πει να μειωθεί η δίκαιη επιστροφή μας θα έχετε τότε περισσότερες δαπάνες. Αυτό μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο όταν θα περάσει το τσουνάμι αυτό της οικονομικής κρίσης και όπου όλοι προσπαθούν να μειώσουν τις εισφορές τους δύσκολα θα μπορέσω να αποδείξω τα πράγματα αυτά στους ψηφοφόρους μου. Γεια. Χάοκ, ναι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή ενημέρωση που μας κάνατε μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έπρεπε να τηρήσετε. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι είναι οι έξι πόροι, οι πηγές πόρων που ψάχνουμε να βρούμε. Ε, ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις, κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη είναι ότι το προφίλ που δώσατε για την νέα αυτή πηγή ιδίων πόρων είναι ε, πάρα πολύ φιλόδοξο εύχομαι καλή επιτυχία και πράγματι να τον βρείτε κύριε επίτροπε γιατί είναι ιδανικός. Ε, θα ήθελα να κάνω μια δεύτερη επισήμανση. Ε, έχετε κατά νου αυτή την περίοδο και για πολλή περίοδο ακόμα θα περάσουμε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη δεν έχει ίδιους πόρους στην ενέργεια, εισάγει και όλη η εισαγωγή της λίγο πολύ ή είναι εχθρικοί προς την Ευρώπη ή πάψανε να υπάρχουν με την αναταραχή που βλέπουμε στη Βόρειο Αφρική. Θα ήθελα αυτό κύριε Επίτροπε να ληφθεί υπόψη γιατί αν επιβαρύνουμε την ενέργεια περισσότερο από ό,τι την έχει επιβαρύνει η Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο στον πλανήτη τότε όλα μας τα προϊόντα και τα αγαθά θα ανατιμηθούν. Γι' αυτό προσέξτε λίγο τον τομέα της ενέργειας στην εξέβρεση αυτής της νέας πηγής ιδίων πόρων. Ευχαριστώ. Τώρα, ένας από αυτούς που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους ιδίους πόρους, ο κ. Λαμασούρ, Ευχαριστώ και τον Γιάννους για τις προτάσεις του καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με τόσο θάρρος δεσμεύτηκε να ε, υποβάλει ε, προτάσεις μέχρι τον Ιούνιο. Μία παρατήρηση και μία σύσταση. Η παρατήρηση έχει ως εξής. Το ψήφισμα που ενέκρινε το Μάρτιο 2007 η Ευρωβουλή περιλάμβανε έξι κατευθυντήρες γραμμές πολιτικού χαρακτήρα που εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα και που νομίζω πρέπει κανείς να τις υπενθυμίζει συνεχώς. Διατήρηση της δημοσιονομικής κυριαρχίας των χωρών μελών, διατήρηση της οροφής των, ε, των ε, ιδιών πόρων, διατήρηση της ουδετερότητας, μείωση των εθνικών εισφορών σταδιακά και εφόσον θα μπαίνουν ε, στο παιχνίδι οι νέοι πόροι, διαφάνεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη και η διασύνδεση της διαπραγμάτευσης ε, πόρος δαπάνη. Εξάλλου, αντίθετα με αυτήν την, ε, με το ψήφισμα του θα ε, είχαν αλλάξει τώρα οι υποψήφοι. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε τώρα τις, το βάρος των προσπαθειών μας. Τώρα, μιλούμε για φόρους, μιλούμε για Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε κρίση αυτά τα πράγματα είναι υπερεκρηκτικά πολιτικά. Πρόκειται για πραγματικά υλικά σχάσεις. Εάν τα χειριστούμε αδέξια θα σκάσουν στα χέρια μας και θα μας σκοτώσουν όλους. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτή την θα έλεγα πυρηνική ενέργεια που έχουμε στα χέρια μας ώστε να παράγει ενέργεια σταδιακά και να μην εκραγεί. Χρειάζεται λοιπόν και κάποια πράγματα τα οποία θα καθησυχάσουν τα νερά. Και επιμένω λοιπόν ώστε και η δική μας η Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθίσουν να σκεφτούν καλά την συζήτηση αυτή πριν από την επίσημη υποβολή προτάσεων τον Ιούνιο, καθώς επίσης και τη συνέχεια που θα δοθεί στις επίσημες προτάσεις. Γιατί και αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν την έννοια μιας πολιτικής συμφωνίας και για το πώς θα συζητηθούν. Διότι αν αρκεστούμε Κάτι που έγινε και το προηγούμενο καλοκαίρι όταν ο Επίτροπος είχε δώσει στο Διεθνή Τύπο μια συνέντευξη για το θέμα αυτό, διακινδυνεύουμε μια τέτοια έκρηξη όπου θα σταματήσει απότομα η συζήτηση τη στιγμή που άρχισε. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν και ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία για τα οποία έχουμε βάλει αυτό το θέμα της διασύνδεσης πόρων και δαπανών στο τέλος των προσπαθειών της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ πριν μπούμε μετά στην φάση επεξεργασίας της έκθεσης. Νομίζω ήταν σωστό και σκόπιμο αυτό ώστε να μπορέσουμε να τα έχουμε συζητήσει όλα πριν να συζητήσουμε αυτό. Ράιμερ Μπέγκε. Σας ευχαριστώ. Ο Αλάν, Αλάν Λαμασούρ, έθεσε πραγματικά το θέμα όπως πρέπει. Πρέπει να συζητήσουμε την ορθή στρατηγική και να υπενθυμίσουμε σε όλες και όλους ότι η συνθήκη απαιτεί από εμά να συζητήσουμε για ιδίους πόρους και να διαπραγματευτούμε τους ίδιους πόρους, διότι χρηματοδοτούμεθα αποκλειστικά από ιδίους πόρους. Θέλουμε να συνεχίσουμε διαρκώς να παραβιάζουμε τις αρχές της συνθήκης, τότε ας μείνουμε σε ένα ποσοστό ας λάβει το Συμβούλιο αποφάσεις και ας πει λυπούμεθα πολύ, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως άλλωστε είπαμε στην προηγούμενη θητεία στην έκθεση του Αλάλα Μασούρ, πρέπει να φύγουν από τη μέση όλες αυτές οι εκπτώσεις. Αυτός ο φρικτός κατάλογος περιλαμβάνεται στο έγγραφο της ε, γραμματείας που δείχνει πώς έγιναν πραγματικά στα όρια της κοινοτική νομιμότητας. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή, να πάυσουν. Και αν καταλήξουμε σε κάποιες αντισταθμιστικέ λύσεις, διότι ίσω αυτό είναι αναπόφευκτο, θα πρέπει να γίνει με διορθωτικούς μηχανισμούς γενικής ισχύω, όχι με ειδικέ εξαιρεσει, με ειδικέ επιστροφές και ούτω καθεξή, για να ικανοποιηθεί πότε ο ένα και πότε ο άλλο. Σημειώνω ότι ο κύριος Επίτροπος μίλησε περί μιας λύσης του ενός τρίτου. Το σημαντικό ερώτημα είναι θα συνεχίσουμε και θα ζητούμε να γίνουν τα πράγματα αυτά όλα διαμιάς ή θα κάνουμε αυτό που λέγεται learning by doing, δηλαδή προχωρούμε σιγά σιγά και διδασκόμαστε από αυτά που επιτυγχάνουμε. Εκτός από το θέμα των ιδιών πόρων, και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνουμε και μια άλλη συζήτηση για διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς διακυβερνητικής χρηματοδότησης ή πράγματα τέλος πάντων τα οποία δεν εντάσσονται επαρκώς στον κοινοτικό προϋπολογισμό που έχουν όμως σχέση με αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα των 27 χωρών μελών. Πώς θα τα χειριστούμε αυτά στο μέλλον δεν θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτά και πιο διαφανή ώστε να επιτρέπουν μια συνολική επισκόπηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και ένα πράγμα θα θέσω υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί παρενέβη σχετικά η Γιούτα προηγουμένως. Υπάρχει ένα έγγραφο του Φεβρουαρίου 1994 όπου τότε η συγκητή Λάγκες λέει ότι η μονομερής αυτή προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απόφαση του Εδιμβούργου οδηγεί σε μια σταδιακή διάβρωση της αρμοδιότητάς της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει να λάβει υπόψη της ποια όργανα λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ευρωπαϊκή κοινότητα. η από τις επιλογές που υπάρχουν επιτάπητος πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα και όλων των μηχανισμών αυτών και να κάνει διαφανείς μεταρρυθμίσεις, να προτείνει διαφανείς μεταρρυθμίσεις, στη βάση όμως πάντως όλων αυτών που ε, απαιτεί η συνθήκη. Νομίζω ότι έχοντας προσπαθήσει κατ' επανάληψη να προωθήσουμε το θέμα των ιδιών πόρων, βλέπετε ήδη υπάρχουν κάποια σχετικά σε έγγραφο του 1994, να συζητήσουμε όλο το εύρος των επιλογών, αλλά να πιέσουμε το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις να προχωρήσει σε περισσότερη διαφάνεια και δικαιοσύνη των ίδιων πόρων. 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Αλλά έστω, διότι θύμισε και τι είπε ο Χόρτ Λάγκε πριν από τόσα πολλά χρόνια, το 1994. Ορίστε. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αμυντική τακτική σε αυτή τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, διότι νομίζω ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις και η εμπιστοσύνη θα πρέπει να αφορά τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουν ένα καλύτερο πρότυπο από αυτό που είχε αρχικά προταθεί το παρόν πρότυπο που έχουμε δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Αυτό ήδη, προ, προελέχθη. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι οι ίδιοι επικεφαλής των κρατών μελών που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, οι ίδιοι υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισαβόνας που αναφέρεται σε νέους ίδιους πόρους και όπως είπε ο Ράιμερ, θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου και να το θεωρήσουμε σημείο εκκίνησης, αν και ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ως προς το 1 τρίτον του προϋπολογισμού, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι πρόκειται για πολιτικό στοιχείο, δημοσιονομικό. Ποιο είναι το υπόβαθρο αυτού του αριθμητικού στοιχείου ή του ποσοστού. Και αν μιλάτε για αντικατάσταση του ενός τρίτου θα ε, πρόκειτο για συνδυασμό ιδίων πόρων ή θα προβάλλατε μία εναλλακτική λύση, μία επιλογή. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θα σήμαινε. Ευχαριστώ που θέσατε και πάλι, που θίξατε και πάλι το γεγονός ότι οι ίδιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι αυτοί και αυτές τώρα που δεν δείχνουν διάθεση να την εφαρμόσουν και ιδίω ό,τι αφορά το δημοσιονομικό της μέρος. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που είπα πριν, ότι το πλεονέκτημα έχει αυτός που ξέρει ανάγνωση. Ορισμένες φορές νομίζω ότι δεν έχουν καν αναγνώσει το κείμενο που υπέγραψαν οι αρχικά των κυβερνήσεων. Ζωζή Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από τις παρεμβάσεις που άκουσα, θα ήθελα να πω ότι δεν θα φτάσουμε σε μία συμφωνία. Γιατί αναφερόμαστε στο άρθρο 311, αναφέρομαι στο άρθρο 311 που προαπαιτεί ομοφωνία για οποιαδήποτε λήψη απόφασης. Άρα δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Θα Υπάρχει κάποιος ίδιος πόρος που θα μπορέσει να εισπράξει άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιο θεσμικό όργανο. Και ποιος θα είναι αυτός ο ίδιος πόρος. Και εάν δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, θα μιλάμε για νέους ίδιους πόρους, δηλαδή για εθνικές εισφορές. Εάν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συλλέξουν τους ίδιους πόρους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μιλάμε στην ουσία για εθνικούς πόρους που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Επίσης, για να υπάρχει καλύτερη αποδοχή από τον πολίτη, δεν θα ήταν σκόπιμο στα πλαίσια των φόρων ή του φόρου διοξιδίου του άνθρακα δεν θα πρέπει να βασιστούμε στη στρατηγική 2020 ή 2020 παύλα 20. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ε, χρησιμότητα αυτού του μηχανισμού, ο οποίος θα πρέπει να γίνει κατανοητός αμεσότερα στον πολίτη. Η συντόνια. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι διότι σήμερα γίνεται αυτή η συζήτηση και χαίρομαι, χαίρομαι διότι συνεχίζεται. Πάντα μου κάνει εντύπωση, μεγάλη εντύπωση ο Αλέν Λαμασούρ που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο οποίος στην ουσία είναι ένας φιλόσοφος των δημοσιονομικών. Πρόκειται για οραματιστές. Εγώ δεν είμαι οραματίστρια, δεν μπορώ να κάνω μια προβολή στο μέλλον και δεν μπορώ να δω να προβλέψω πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2014. Δεν θέλω βεβαίως να φανώ απεσιόδοξη, δεν είναι αυτός ο στόχος μου, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει συνεχώς να βλέπουμε την πλευρά των εσόδων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για το από πού προέρχονται τα χρήματα. Η συζήτηση είναι άκρο σημαντική. Όμως, ελέγχθη σαφώς ότι η συζήτηση ακολουθεί μία περίοδο κλειδονισμών. Τώρα έχουμε φτάσει σε μία ιδιαίτερα ζωηρή συζήτηση, αλλά θα ήταν ε, λυπηρό αν ε, κάνουμε έναν άμεσο συσχετισμό με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο των ιδίων πόρων. Γιατί θα πρέπει να εργαστούμε με το τρέχον σύστημα για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα συζητήθηκαν επί μακρόν, αλλά υπάρχουν και πλεονεκτήματα. Δεν χρειαζόμαστε ένα ειδικό σύστημα συλλογής ίσπραξης φόρων, άρα υπάρχει ένα εύκολο πλαίσιο, ένα ε, πλαίσιο εύκολης ίσπραξης. Ως προς την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η αρχή, θα πρέπει να την σεβαστούμε και πίσω να έχουμε επιπρόσθετους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια ενός ενωτικού ε, πλαισίου. Δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά έσοδα για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα της ενότητας του προϋπολογισμού. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η αρχή και Θα πρέπει έτσι να τροφοδοτείται ολόκληρος ο προϋπολογισμός και όχι επιμερισμένα. Το έχω ανάψει τώρα, λέει η Ιούτα. Μέχρι τώρα όμως δεν την ακούγαμε. Ελπίζω, λοιπόν, εφόσον ε, προχωρήσεις πιο βαθιά στην συζήτηση να έχεις και περισσότερο θάρρος για να μιλήσεις και με τα τμήματα εκείνα του Συμβουλίου που στέκονται ακόμα απολύτω αρνητικά απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος ιδίων πόρων. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ιδίων πόρων που να είναι πιο διαφανές, πιο δίκαιο και που παρόλα αυτά να προσφέρει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τα χρήματα που χρειάζεται για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Δεν τις έχουμε αναλάβει μόνοι μας, μαζί με το Συμβούλιο τις έχουμε αναλάβει. Παρακαλώ λοιπόν δείξτε λίγο περισσότερο θάρρος. Μην είμαστε τόσο ταπεινόφρονες. Γνωρίζω ότι χρειάζεται και πολλή δουλειά και πολύ πειθό όχι μόνο απέναντι στο Συμβούλιο, αλλά και απέναντι και σε όλες και όλους τους συναδέλφους μας και βεβαίως και απέναντι στην κοινή γνώμη. Αλλά πρέπει τουλάχιστον τώρα να δείξουμε το θάρρος αυτό, όπου καλούμαστε να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κοινό που θα θαυμάζει με τα μάτια ανοιχτά από το 2014 και μετά ένα νέο μηχανισμό. Ο Επίτροπος τώρα για απαντήσεις στον τελευταίο αυτό γύρο των απαντήσεων, αλλά παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο, διότι στο τέλος θέλουμε να δώσουμε άλλα πέντε λεπτά στον εισηγητή μας. Καλά τα πάμε ακόμη από χρόνο, αλλά να το πάμε μέχρι τέλους καλά. Θα μπορούσε και να απόσχω, λέει ο κ. Λεβαντόσκη, και να πάρει αμέσως τον λόγο ο Σαλβατόρ Καρίγα και να μιλήσει για περισσότερο από πέντε λεπτά. Τώρα, κύριε Βόγκαν, άκουσα πραγματικά από τα χείλη σας ε, τις απόψεις των ευρωσκεπτικιστών. Υπό ορισμένες συνθήκες υπάρχει η δυνατότητα τώρα να ανοίξει το θέμα των ιδιών πόρων και η πραγματική δεξιότητα θα είναι, θα έγκυται στο να διατηρηθεί ανοιχτό το θέμα και να μην κλείσει αμέσω. Μέχρι ότου να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το James Ellis ε, ρώτησε σχετικά με την τεχνητή μείωση του ε, ΦΠΑ που νομίζω ότι έχει φτάσει τώρα στο 0,3%. Πάντως είναι ένα σύστημα επιβαρημένο με πολλές εξαιρέσεις. Η Γερμανία έχει μειώσει ακόμη περισσότερο, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι στο 0,1% 10% από το αρχικό. Έχουν μειωθεί λοιπόν αυτά. Τώρα πώς να πείσουμε τους Βρετανούς ψηφοφόρους. Ίσως πρέπει να βρεθεί κάποιος αρκετά ικανός και ανταγωνιζόμενος στον τύπο του Ρούπερτ Πέρντοχ ώστε να μπορέσει να τους πείσει. Για παράδειγμα να μιλήσει στους Ουαλούς που ε, απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Ορισμένοι εξ αυτών, οι Κορνουάλοι για παράδειγμα, δείχνουν και υποστήριξη. Αλλά βέβαια σε άλλα τμήματα της χώρας σας είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ε, βέβαια προστιθέμενη αξία, αλλά αυτό είναι λίγο και σύνθημα. Βλέπουμε όμως και αυτό το pooling πόρων, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το κανάλι της μάχης που ε, κάνει βέβαια πιο δύσκολη την χρήση ή την ολοκλήρωση διευρωπαϊκών ε, δικτύων. Όσο, για να αφορά, όσον αφορά το call rate αυτού του ΦΠΑ, αυτή είναι η εξήγηση. Ότι ένα κλάσμα μόνο ε, παραμένει. Γιατί κυρία Τζαβέλα, ναι, αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη τώρα είναι δουλειές και απασχόληση και μελέτη επιπτώσεων για οποιοδήποτε θέμα είναι σημαντική. Η ενέργεια, η, ενδεχόμενα δηλαδή οι ήδη πόροι από την ενέργεια θα είναι μάλλον για να βουλώνουν κάποιες τρύπε και δεν θα επιβάλλουν τόσο μεγάλο βάρος στην φορολόγηση. Για τον αλλά συζητώντας ιδίους πόρους παρόντος το Αλάν Λαμασούρ είναι σαν να προσπαθώ να παίξω πιάνο παρόντος του Φρέντερικ Σοπάν. επαναλάβατε τις βασικές αρχές και ο Ράιμερ Μπέγκε το ίδιο και η Ελγκα το ίδιο για θέματα επικοινωνίας για την διατήρηση ανοιχτού του θέματος δηλαδή μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και εδώ πρόκειται άλλωστε περί επικοινωνίας πριν από την ανακοίνωσή μας δηλαδή για την απόφαση για τους ίδιους πόρους. Μιλούμε πλέον ουσιαστικά για εβδομάδες και μήνες. Τις επιλογές μας πρέπει να τις οριστικοποιήσουμε στην Κομισιόν τα τέλη Μαρτίου και είναι ασφαλώς και πολύ σημαντική η επικοινωνία καθώς και η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2012 που θα προκαλέσει άλλο γύρο συζητήσεων γύρω από την Ευρώπη. Για τον Ράιμερ αυτή η ιδέα της σταδιακής εφαρμογής του facing in των ιδίων πόρων δεν αποκλείεται. Δηλαδή να πάμε σιγά σιγά σε αυτούς τους ίδιους πόρους και όχι να πηδήξουμε ε, στα νερά μια και καλή. Δηλαδή αυτό που μου αρέσει είναι αυτό το αγγλικό up to, μέχρι. Ποσοτικοποιώντας έτσι τις φιλοδοξίες μας. Θα πρόκειται για συνδυασμό ιδίων πόρων. και όχι επιλογή ενός νικητού των, μεταξύ των υποψηφίων. Εγώ είμαι από τη γενιά της αλληλεγγύης και είπαμε θάρρος αλλά και σοφροσύνη. Γι' αυτό και καταφέραμε να κάνουμε ανέμακτη επανάσταση και ελπίζω να μην υπάρξουν και άλλα, θέματα, άλλα θύματα μάλλον στην πορεία μας προς τις ε, νέες, ε, προς νέους ίδιους πόρους. Ενώ η Σιδονία που είναι ε, από τη γενιά μετά την γενιά της αλληλεγγύης είναι λιγότερο αισιόδοξη. Κύριε Φερνάντες, επανέλαβα όλες τις αρχές. Πρόκειται να χτίσουμε ένα σύστημα και για την επικοινωνία δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες. Να έχει όμως διαμεθοριακό χαρακτήρα. Είναι πιο εύκολο να πάμε κατευθείαν στις Βρυξέλλες και όχι μέσω των εθνικών φυσαυροφυλακίων να υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο μόνο τα εισφορές από την τις ε, αεροπορικές μεταφορές και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ε, και τα λοιπά μπορούν να λειτουργήσουν στο επίπεδο αυτό. Όλα τα άλλα θα πρέπει να έχουν κάποιο ενδιάμεσο στάδιο, το οποίο βέβαια δεν είναι πλέον έκτημα για την Σιδωνία, ναι, περισσότερο θάρρος. Ας μην θυμόμαστε τις ρομαντικές εποχές ε, της αλληλεγγύης, Ποιο θα φανταζόταν τότε ότι θα έμπαινε μια κυρίαρχη Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, Γιάννου, σωστά, αλλά λέει η Γιούτα Χάουκ. Α, αμέσως, αμέσως. Πρώτα χειροκρότημα. Μπορούμε να χειροκροτήσουμε και τους λιγότερο ταλαντούχους πιανίστες, αλλά βέβαια οι λιγότεροι ταλαντούχοι πιανίστες θα κάνουν ε, θα επιτελέσουν πρόοδο μόνο εφόσον βρίσκουν και αναγνώριση των προσπαθειών τους ε, πει προσωπικού το, τα, η φιλοφρόνηση που έκανε για μένα δεν προσθέτει τίποτε στην δόξα του Σοπέν και μάλλον θέτει σε κίνδυνο την συνέχεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας διότι μας βλέπουν και με το web stream τώρα πια όλος ο κόσμος θα θεωρεί ότι είμαι ο Σοπέν της φορολογίας αυτό μου φαίνεται ότι είναι βαρύ πλήγμα Σωστά. Σαλβαδόρ, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος μετά από αυτή τη μουσική παρεκτροπή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο για την αποκαλυπτική του εισήγηση για το πώς έχει η κατάσταση. Πρόκειται για θέμα θάρρους. Θα πρέπει όλοι να δείξουμε περισσότερο θάρρος, αλλά είναι αυτό πολλές ε, δύσκολο όταν ξέρουμε ότι ε, ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι όταν προβάλλουμε ορισμένες λύσεις. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για φορολόγηση, για εισφορές και ιδιαίτερα για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ίσως το Συμβούλιο να αντιδράσει και να καταπνίξει αυτή την προσπάθεια εν τη γενέση της. Από την άλλη πλευρά, για να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα από το παρόν, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι, δηλαδή να μην αλλάξουμε άρδιν το σύστημα ιδίων πόρων, να προβάλλουμε μία κλιμακωτή τροποποίηση. Όμως Υπάρχουν λόγοι για, τη, για τους οποίους αυτός ο τέταρτος πόρος μετατράπηκε στον σημαντικότερο πόρο και τον ε, μοναδικό δημοσιονομικό πόρο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις εισφορές ε, βάση του ΑΕΠ. Μιλούσαμε για ένα συμπλήρωμα πόρου Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν έφτασε σε αίσιο πέρας. Αυτός ο τέταρτος πόρος αποτελεί ένα νέο σύστημα ίσπραξης. Υπάρχει ίσως γενική συνένεση ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει, αλλά με βάση ποιες αρχές αντικατάσταση της παρούσας χρηματοδότησης ή προσθετικότητα, συμπληρωματικότητα ή να αλλάξουμε τη σύνθεση των ε, δημοσιονομικών εσόδων ή να συμπληρώσουμε αυτούς τους πόρους με νέους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ε, πόρους, αλλά έναν καλύτερο ε, τρόπο επιβολής ε, φορολόγησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα ίσπραξης. Αν πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό, εάν δεν μπορέσουμε να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα την Επιτροπή, ως το θεσμικό όργανο που θα προβεί σε αυτή την εισπράξη, τότε θα μιλήσουμε για μεταφορές ή νέες χρηματοδοτήσεις. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτόνομος μηχανισμός ύπαρξης, τότε δεν θα θεωρηθεί από τα κράτη-μέλη ως ε, κοινοτικός αλλά ως εθνικός μηχανισμός. Άρα φτάνουμε στο αρχικό μας σημείο, κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να μιλάμε για καθαρούς εισφορείς και καθαρούς αποδέκτες. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη αυτό το μηχανισμό εισπράξης ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινοτικός και αυτό αυτόνομος. Ως προς το ΦΠΑ, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο ΣΟΥΡ το συζητήσαμε. Θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη το εξής. Οι εθνικές δαπάνες θα πρέπει να θεωρηθούν κοινοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ως προς τις υποδομές, την εξωτερική δράση, τις δράσεις στον τομέα της ενέργειας και όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να μεταφερθούν σε δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει ε, αυτή την αρχή να λάβουμε υπόψη, γιατί μία από τις ε, βασικές ε, πηγές είναι η εξοικονόμηση και η μεταφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Και ως προς τα κριτήρια που είναι σαφή για όλους και που ορίζουν τους νέους ίδιους πόρους. Δεν μιλάμε για μεταφορές από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μιλάμε για διασυνοριακή εισπράξη που να συνδέεται στις, με τις κοινοτικές πολιτικές και να συνδέεται και με την εσωτερική αγορά. Και τέλος, δεν θα πρέπει οι πολίτες να θεωρήσουν ότι πρόκειται για έναν επιπρόσθετο φόρο που θα τους επιβαρύνει επιπροσθέτως. Θα πρέπει να απαλύνουμε αυτό το πλαίσιο με τη μεταφορά, μάλλον τη δημιουργία ενός κοινοτικού καθαρά πόρου. Θα πρέπει να αλλάξω λοιπόν την ε, έκθεσή μου κατά κάποιο τρόπο και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλουν ε, τροπολογίες μέσα στα πλαίσια αυτής της δίμηνης διαδικασίας, έτσι ώστε τον Ιούνιο να έχουμε μια τελική πρόταση, η οποία να βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αποφάσεις της. Σας ευχαριστώ, Σαλαδόν. Θα σου αφαιρέσω και τρία τέταρτα του λεπτού που υπερεύεις. Ναι, καλά, τι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ τώρα ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας ε, συνεδριάσεως. Συζητήσαμε τους ιδίους πόρους με τη στενότερη έννοια και στο δεύτερο μέρος όπου θα μιλήσουμε για καινοτόμα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Καλωσορίζω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, κ. Μάιστατ. Καλώς ήρθατε. Θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Ο Σαλβαδόρ θα λάβει τώρα πλέον 3,5 μόνο λεπτά, αντί των 5 λεπτών, Αστειεύομαι. Θα κάνει την εισαγωγή ο Σαλβαδόρ Γαρίγα μετά 7 λεπτά ο Επίτροπος ή μήπως θέλει οπωσδήποτε 10. Καλά, θα δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε. Μετά ο κύριος Μάιστατ και μετά θα προχωρήσουμε σε γύρο ερωτήσεων με πρώτα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ εντάχει γιατί βλέπω ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, κάτι που δεν ίσχυε πριν. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο είναι πώς θα περιορίσουμε τους πόρους μέσα στα πλαίσια και των επενδύσεων, των εισφορών δηλαδή μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 ε, και των νέων προαπαιτήσεων της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για στοιχεία ύψης της σημασίας διότι έχουμε 126 δις ευρώ σε πιστώσεις δαπανών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο έτος και η Επιτροπή για την εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων όπως τα ΤΕΝ, το ενεργειακό δίκτυο, η μεταρρύθμιση των υποδομών, ε, το δίκτυο το, ε, ε, το ευρυζωνικό οδηγεί σε 2-3 Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε τη διάσταση αυτού του εγχειρήματος, δηλαδή τους ε, πόρους και το τι προαπαιτείται για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη έλλειψη συμμετοχής ε, ιδιωτικών επενδύσεων και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο για τον ε, προϋπολογισμό να δράσει ως καταλήτης των ε, δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Γι' αυτό αποτύχαμε και στις οικονομικές εταιρικές ε, σχέσεις στις ΣΟΕΣ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να λάβουμε υπόψη ότι εδώ και 10 χρόνια στις ε, ε, δημοσιονομικές προοπτικές μιλάμε για 1,3% του προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Και το ελεγκτικό συνέδριο ε, αξιολογεί θετικά αυτό, αυτά τα μέσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μέισταντ και θα ήθελα να τον ρωτήσω τι πιστεύει για την χρήση αυτών των μέσων από πλευρά ΣΕΤΕ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί τους ιδιωτικούς και δημόσιους ε, μηχανισμούς επένδυσης από ένα έως ε, στο 5%, το στο 5% και η ΕΤΕ πολλαπλασιάζει επί τέσσερα το, τις δανειοδοτήσεις μέσα στα πλαίσια αυτής της δεκαετίας και μιλάμε για 800 δις ε, τελικά, κάτι το οποίο δεν είναι κατώτερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μάιστατ, τι πιστεύεστε για τις δαπάνες που προβλέπονται μέσα στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Πώς μπορούν να καλυφθούν από τα νέα χρηματοοικονομικά μέσα ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας και των μεταφορών. Ε, βεβαίως υπάρχουν ε, και άλλοι τομείς που χρήζουν επενδύσεων, τα διαρθρωτικά ταμεία και η ΕΤΕ θα μπορέσει να δράσει περισσότερο, διότι βοηθά στην συγχρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη-μέλη. Μπορούν να δοθούν και προκαταβολές δηλαδή πώς θα αξιολογήσουμε αυτά τα νέα δημοσιονομικά μέσα με τον δημοσιονομικό κανονισμό που τώρα αναθεωρούμε. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό σε αυτά τα νέα μέσα. Και όπως είδαμε από τον τύπο, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα ευρωομόλογα, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον ε, πρόεδρο της ΕΤΕ πώς ε, λειτουργούν αυτά τα ευρωομόλογα και πώς θα δράσει η ΕΤΕ και ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των νέων Eurobonds και του κινδύνου που θα πρέπει να αναλάβει κανείς μέσα στα πλαίσια δημιουργίας εγγυήσεων, κατάλληλων εγγυήσεων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε αυτό το συσχετισμό ε, κινδύνου και πολλαπλασιαστικού ε, δίκτυ. Αυτά θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εσείς τώρα, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστώ και σας Σαλβαδόρ που θέσατε τις περισσότερες ερωτήσεις ήδη στον Πρόεδρο κύριο Μάιστατ. Έτσι εγώ θα μιλήσω λιγότερο με την αδειά σας. Η πρώτη δήλωση για τους ιδίους πόρους η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε την ε, δημοσιονομική κυριαρχία των χωρών μελών. Για τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα πρέπει αυτά να συγχέονται με τα ευρωομόλογα, διότι εφόσον υπάρχει τέτοια σύγχυση, αμέσως προκαλούμε αντιδράσεις ορισμένων χωρών μελών που φοβούνται ότι θα χρεωθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το τελείως διαφορετικό. Πρόκειται όμως για καινοτόμα μέσα τόνωση των επενδύσεων, κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων, και με σημαντικό ρόλο βέβαια και της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων, αν και όχι μόνο. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα ήδη λειτουργούν. Ήδη υπάρχουν για την περίοδο 2007-2013 οι μείζονες τομείς λειτουργίας τους είναι για μεγαλύτερους όγκους, για παράδειγμα για καταμερισμό των ε, κινδύνων, ένα δισεκατομμύριο για την έρευνα, επίσης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, μισό δισεκατομμύριο, επίσης για, ε, για το επιχειρήν, προσφέροντας χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μέχρι τώρα εφαρμογές και είναι βέβαια και ένα πεδίο συλλογής εμπειριών για να μπορέσει να προσφερθεί ακόμα μεγαλύτερη ε, τόνωση μετά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου ε, χρησιμοποιούνται αυτά. Δεν θα μπω όμως αυτή τη στιγμή σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά είναι σαφές ότι μετά το 2013 θα πρέπει να έχουμε περισσότερα τέτοια καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, διότι έχουμε κάποιους περιορισμούς από τον προϋπολογισμό και έχουμε και ξεκάθαρα ορισμένα κενά στις υποδομές μεταφοράς ενέργειας. Ε, εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο ομόλογα ευρωπαϊκών έργων που για τα αυτά μίλησε ο πρόεδρος Μπαρόσο στην ομιλία του περί της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και έχουμε βάλει στο δημοσιονομικό κανονισμό ένα τμήμα για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Ναι, ναι, είστε και έτοιμοι να επικρίνετε βεβαίως. Ως ό,τι αφορά τις αρχές, καλύτερα να τα συζητήσει ο ίδιος ο πρόεδρος ε, Μέιστατ, αλλά αυτό που ε, οι βασικές αρχές είναι απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος, όχι να υπάρχει ένα μέρος του προϋπολογισμού που να είναι εκτός ελέγχου. Εμείς είμαστε υπέρ του streamlining, υπέρ μιας τυποποίησης των ε, χρηματοδοτικών μέσων που αυτή τη στιγμή γίνονται περισσότερο ad hoc και επίσης τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν μπορούν παρά να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δοθέντων των περιορισμών και όπως είπα θα μπορούσαν ε, να προβλεφθούν μέχρι το 2014. Ο κύριος Πόρτας είναι έτοιμος να με κατακεραυνώσει. Όχι, βλέπω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Γιούτα Χάουκ, σας ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Πιστεύω ότι υπάρχουν ε, τρία σημαντικά στοιχεία τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά. Καταρχάς, ο εισηγητής σας το είπε, τεράστιες ανάγκες επενδυτικέ έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Ο εισηγητή σας ε, αναφέρθηκε σε μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τι ανάγκε επενδύσεων. Αν θέλουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020, οι επενδύσεις αντιστοιχούν σε 3.000 δισεκατομμύρια 3-3 ευρώ μόνο και μόνο για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το το δίκτυο, το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών χρειαζόμαστε ένα τεράστιο ποσό μέχρι το 2020, επομένω τεράστιες επενδυτικές ανάγκες. Ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι οποίοι δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Οι εθνικοί προπολογισμοί για τα περισσότερα κράτη-μέλη βρίσκονται σε μία φάση δυσνομική εξυγίανση και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάζομαι εδώ πέρα που πιστεύουν ότι θα υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στον κοινοτικό προπολογισμό. Άρα έχουμε και δημοσιονομικούς προορισμούς. Τρίτον, η χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα θα παραμείνει περιορισμένη, ιδίως όσον αφορά τον, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ξέρετε ότι ο τραπεζικός τομέας δεν έχει εξηγιανθεί εντελώς οι νέοι κανόνες επιτήρησης της Βασιλείας 3, που είναι δικαιολογημένοι βέβαια, θα έχουν όμως και μια επίπτωση όσον αφορά τον, τη χρηματοδότηση, τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τον δανεισμό. Επομένως, πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε ένα κάποιο τρόπο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις επενδύσεις, έχοντας λιγότερα μέσα ή τα ίδια τουλάχιστον δημοσιονομικά μέσα. Βάσει λοιπόν αυτών συζητάμε τα συνδυασμένα αυτά χρηματοδοτικά μέσα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για να συνεχίσουμε με το μουσικό αυτό παράδειγμα θα πρέπει να παίξουμε πιάνο με τέσσερα χέρια, μόνο και μόνο για να καταφέρουμε να αυξήσουμε τον ήχο τελικά. Έχουμε όμως ήδη μια κάποια εμπειρία για τα συνδυασμένα αυτά μέσα. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα μέσα αυτά και για ποια σχέδια. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία έχουν εσωτερικό ποσοστό επιστροφής των επενδύσεων πολύ χαμηλό και πολλές φορές αρνητικό. Πρόκειται για έργα όμως τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά από οικονομικής πλευράς. Όμως το ποσοστό επιστροφής των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλό. Γι' αυτά καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστούμε και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει λοιπόν να καταργηθούν αυτές οι επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προπολογισμό για τα συγκεκριμένα αυτά έργα. Από την άλλη έχουμε έργα τα οποία έχουν ποσοστό εσωτερικής απόδοσης πολύ πιο υψηλό. Έργα με μικρότερο κίνδυνο αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εμπορικέ τράπεζες. Μεταξύ των δύο αυτών άκρων όμω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία έχουν μια κάποια αποδοτικότητα περιορισμένη, τα οποία έχουν ένα ψηλό επίπεδο κινδύνου, έργα τα οποία δεν μπορούμε να προτείνουμε αν θέλετε στις τράπεζες που δεν θα μπορούσαν εύκολα να αποδεχθούν οι τράπεζες για δανεισμό. Ανάμεσα στα έργα αυτά έχουμε αρκετά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση, είναι σημαντικά για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Γι' αυτά ακριβώ λοιπόν τα έργα τα οποία βλέπετε και στη διαφάνεια, τα οποία βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα, στο μεσαίο τμήμα τη διαφάνεια αυτή, γι' αυτά τα έργα πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε κοινά συνδυασμένα μέσα χρηματοδότηση. Γιατί με λίγα χρήματα από τον κοινοτικό προπολογισμό θα καταφέρουμε να έχουμε ένα φαινόμενο μόχλευση, θα καταφέρουμε ουσιαστικά να αυξήσουμε την επενδυτική του ελκυστικότητα και κατά αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε περισσότερο το δανεισμό από τι τράπεζε. Έχουμε το Τζέσικα, τον Τζάσπερ, το Τζέρεμι όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε έναν μηχανισμό που ονομάζεται RSFF, μηχανισμός χρηματοδότησης με, με επιμερισμό των κινδύνων όσον αφορά την έρευνα. Και έχουμε επίσης ένα μηχανισμό LGTT, μηχανισμός εγγύησης δανείων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Καλύπτουμε εδώ πέρα λοιπόν μέσω εγγύσεων ένα πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο. Τον κίνδυνο ο οποίο εμφανίζεται τα πρώτα χρόνια κατασκευής υλοποίησης συγκεκριμένων έργων. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συνδυασμένα μέσα χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων για την έρευνα μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει δάνεια για 6 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την έρευνα και το κόστος για τον κοινοτικό προπολογισμό είναι 390 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με μικρό ποσοστό του κοινοτικού προπολογισμού καταφέρουμε να έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο πιο ελκυστικό το συγκεκριμένο έργο και μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Όσον αφορά το μηχανισμό εγγύησης δανείων για την ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θέλετε, όλη η εμπειρία το όλο εγχείρημα, αλλά χάρη στο μηχανισμό αυτό καταφέραμε να προσελκύσουμε επενδύσεις ε, για τον τομέα των μεταφορών για 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ με κόστος 140 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον κοινοτικό προπολογισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο της μόχλευσης διαφέρει προφανώς από τον έργο στο άλλο, πάντως υφίσταται και είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αφού του είδους τα κοινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μείνουμε σε κάποιες αρχές, η αρχή της Απλότητα ε, καταρχής τη απλούστευση, Δεν θα πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα χωρίς λόγο. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες, απλές, ευκολοκατανόητες από τους χρήστες και πιο ορατές επομένως για τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεύτερη αρχή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος revolving, δηλαδή δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης κάποιων ταμείων, κάποιων πόρων, ακριβώς επειδή θα υπάρχει αυτό το πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Αν καταφέρουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ένα πολλαπλασιασμό της απόδοσης των επενδύσεών μας, τα νέα αυτά χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν άλλες επενδύσεις. Και τέλος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, και τις δυνατότητες που μας δίνονται για να προσελκύσουμε επενδύσεις από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εργάζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια μάλιστα τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται στον έλεγχο του λεκτικού συνεδρίου κάθε φορά που χρησιμοποιεί ακόμα και ένα ευρώ μόνο από τον κοινοτικό προπολογισμό. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα ζητήσουμε καμία εμεί ε, εξοδότηση χωρί έλεγχο. Αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιούμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα χρησιμοποιεί έστω και περιορισμένο ποσό από το κοινοτικό προπολογισμό, αυτόματα θα ξεκινάει και το σύστημα ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο. Για να σεβαστώ και το χρόνο που μου έχει δοθεί, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του εισηγητή σας για τα project bonds, τα euro project bonds. Ο πρόεδρος Μπαρόζο όντω είναι αυτός ο οποίος παρουσίασε πρώτος την ιδέα αυτή και όπως πολύ σωστά είπε ο επίτροπο Λεβαντόσκι, δεν έχει καμία σχέση αυτό το Euro Project Bond με τα περίφημα ευρωμόλογα για τα οποία μιλάμε πολύ τελευταία. Αυτοί που μιλάνε για ευρωομόλογα ουσιαστικά μιλάνε για ομολογιακά δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. Εδώ αναφερόμαστε καταρχάς σε ομολογιακά δάνεια που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένου οικονομικού φορεί που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα. Ποια είναι η βασική ιδέα. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών που υπάρχουν, θέλουμε να προσελκύσουμε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ασφαλιστικούς οργανισμούς, από pension funds, από ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, από οργανισμούς που μπορούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. Αυτοί όμως μπορούν να δανείσουν, να επενδύσουν μέσω συγκεκριμένων ομολογιακών δανείων ενός κάποιου επίπεδου, δηλαδή να έχουν μια βαθμολόγηση α ή διπλό α. Επομένως, ο μηχανισμός των Euro Project Bonds μας επιτρέπει να συνάπτουμε ομολογιακά δάνεια, ομόλογα, τα οποία θα βασίζονται, που μάλλον αν βασίζονταν μόνο στο επίπεδο, στην ποιότητα του project, θα είχαν μια βαθμολογία Β ή διπλό Β. Θέλουμε να αυξήσουμε τη βαθμολόγηση αυτή στο Α ή στο διπλό Α, αυξάνοντας το τμήμα του δανείου, το οποίο ονομάζεται senior debt, δηλαδή το κύριο αυτό χρέος, με την χρησιμοποίηση ενός ε, άλλου τμήματος του χρέους, το οποίο ονομάζεται Junior debt υπαγόμενο χρέος. Εκεί ακριβώς επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δημιουργώντας αυτό το επίπεδο, αυτό το τη στρώση του junior debt, του υπαγόμενου, χρέ, υπαγόμενου χρέους, χρέος υπαγόμενου για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυξάνεται αυτόματα η ποιότητα του, της άλλης σα του δανείου, της άλλης Συνιστόσα του χρέους που ονομάζεται senior debt του κυρίου χρέους δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει ένα χρηματικό ποσό από τον προπολογισμό για να δώσει μία πρώτη εγγύηση. Το σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι σε κάθε περίπτωση η δέσμευση του κοινοτικού προπολογισμού θα είναι περιορισμένη από την αρχή. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν θα δημιουργηθεί μία πολύ μεγάλη αχαλήνοτη ευθύνη. Ήδη από την αρχή θα γνωρίζουμε ποια είναι η εγγύηση την οποία φέρει ο κοινοτικό προπολογισμό. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τουλάχιστον θα έχει χαθεί μόνο αν θέλετε το αρχικό αυτό ποσό, αλλά στι περισσότερε περιπτώσει, και αν έχουμε επιλέξει καλά τα έργα, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εξ αρχή λοιπόν το ποσό αυτό από τον κοινοτικό προπολογισμό θα έχει ένα περιορισμό, ένα πλαφόν. Το υπολοιπόμενο κίνδυνο θα τον αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εμείς να λάβουμε την επιπλέον ευθύνη, την επιπλέον εγγύηση. Αυτή είναι η βασική ιδέα των Euro Project Bonds. Πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε επενδύσει από τον ιδιωτικό τομέα για σημαντικά έργα υποδομή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προς Θεού θέλει μάλιστα και με τέσσερα χέρια να παίξει πιάνο ο Πρόεδρος με τόσους πιανίστες και τόσο αριστοτέχνες εγώ αναγκαστικά θα χρειαστεί να προσθέσω άλλο όργανο στη συζήτησή μας, δηλαδή το τύμπανο. Το τύμπανο για να κάνουμε θόρυβο και να προσελκύσουμε την προσοχή στα επιχειρήματά μας. Φρανκ Έγγελ είναι ο πρώτος ωστόσο που θα αναλάβει να μιλήσει όλα αυτά μας οδηγούν σε μία μορφή εφωνίας ή πολυφωνίας. Την επόμενη φορά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεδριάσουμε σε ένα οντιτόριουμ διότι οι μουσικές μας φιλοδοξίες δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλο έδαφος εδώ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για καινοτόμα δημοσιονομικά σχέδια. Την ε, τελευταία φορά που μιλήσαμε, μάλλον την πρώτη φορά που έγινε λόγος για σχέδιο, ε, για σχέδιο συνθήκης το 53, είχε γίνει λόγος για ε, η οικονομική κοινότητα η οποία θα συνάψει συγκεκριμένα δάνεια Είτε μιλούσαμε για project bond, είτε για eurobonds. Εδώ, για, για, εδώ και 57 χρόνια βλέπουμε ότι χρειάζονται χρηματοοικονομικά μέσα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εδώ έγκυται και η δυσκολία διότι τα κράτη-μέλη παλινοδούν, δεν θέλουν να δώσουν περισσότερο χώρο στην Ένωση και βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με αριθμητικά στοιχεία που αποκλίνουν. Θυμάμαι ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ στην ε, Επιτροπή μας είχε πει ότι οι δικές του εκτιμήσεις για τον ε, δικό του τομέα, δηλαδή για τα ενεργειακά δίκτυα και τα σχετικά μέχρι το 2020, αποτελούν μία ε, επένδυση μια επένδυση της τάξης των 2 δις ευρώ. 2-3 με συγχωρείτε ευρώ. Ή 3-3. Για την ε, στρατηγική του 2020. Αυτό αφορά πολύ υψηλά ποσά. Εάν μιλάμε για 2-3... Μιλάμε για 200 δις ετησίως. Άρα μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση μόνο με το γεωργικό τομέα. Το πρόβλημα αρχής, το θέμα αρχής έγκυται στο εξής. Θα έχουμε να κάνουμε με ένα πολλαπλασιαστικό ε, σχήμα το οποίο θα βρίσκεται εκτός ελέγχου. Άρα, αργά ή γρήγορα θα μιλάμε για θέμα δημοκρατικής νομιμότητας. Καταλαβαίνω τους λόγους ε, του, της ύπαρξης του εγχειρήματος, όμως υπάρχει μεγάλη οξύτητα ως προς το θέμα της λογοδοσίας που θα φυγεί αργά ή γρήγορα. Βεβαίως δρούμε κατά αυτό τον τρόπο, διότι μερικοί αντιτίθενται σε αυτές τις ε, αυξήσεις, αλλά δεν αντιτίθενται για αυξήσεις ως προς πολιτικές που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν. Ως προς τα project bonds τώρα, Για λόγους πατριωτισμού αλλά και λογικής θα προτιμούσα να μιλήσουμε ε, μέσα σε ένα λελογισμένο πλαίσιο όπου το, τα επιτόκια θα ήταν χαμηλότερα από οπουδήποτε αλλού μέσα στα πλαίσια αυτού του κυκλώματος, του δημοσιονομικού κυκλώματος και μέσα στα πλαίσια της ε, ρευστότητας της αγοράς. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ταξινομήσουμε τα Eurobonds με τα Project Bonds τώρα που μας έθιξε ο κύριος Μεϊστάτ θα δεχόμασταν ένα υψηλότερο ε, θα υπήρχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τα Eurobonds σε σχέση με το suboptimal, μια suboptimal προσέγγιση και θα ήθελα να την ξανασκεφτούμε. Για να μην μιλάμε για υψηλότερο bond. Ε, επειδή καταρχήν θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το δεχτούμε ή όχι. Σας ευχαριστώ κάπως ε, περισσότερο, κάπως ε, ξεπεράσατε το χρόνο σας. Εσείς τώρα, κύριε Καλφίν, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μάιστατ για την εξήγηση του θεού για την παρουσίαση του θέματος. Τα όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων είναι θετικά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τριών ειδών εμπλοκές και έξτρα χρηματοδότηση από τα χρηματοδοτικά όργανα για έργα τα οποία είναι εμπορικά βιώσιμα αλλά χρειάζονται σημαντική πρώτη επένδυση upfront και εδώ και η τράπεζα αλλά και άλλα ίσως ε, ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν αυτή τη χρηματοδότηση μέχρι ότου να μπουν μέσα οι υπόλοιποι επενδυτές. Δεύτερη περίπτωση είναι όταν θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και άλλα πιστοτικά ιδρύματα να καλύψουν μέρος του κινδύνου έτσι ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα για τους ε, ιδιώτες επενδυτές. Λίγο πολύ αυτό είναι και αυτά τα European Project Bonds που ε, εξήγησε ο πρόεδρος Πάιστατ. Και ε, ο τρίτο, το τρίτο είδος χρηματοδοτήσεως που προσεγγίζει πολύ περισσότερο σε επιδοτήσεις και χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι έργων που, όπου δεν καλύπτεται μόνο ο κίνδυνος αλλά υπάρχει και συμμετοχή ε, δημόσιας χρηματοδότησης πλέον δοθέντων των μεγεθών, μιλήσαμε για τα μεγέθη της ε, χρηματοδότησης της ενέργειας, αλλά υπάρχουν και άλλες ανάγκες στις μεταφορές, για παράδειγμα. Μιλούμε εν τέλει για τεράστια ποσά χρημάτων. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ιδιωτική επένδυση, να τις προσφερθούν κίνητρα δηλαδή, εάν σκεφτούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόσθετη κάλυψη κινδύνου, και θα πρέπει να υπάρχουν και αρκετά δημόσια χρήματα είτε από τους εθνικούς προπολισμούς είτε από τον ευρωπαϊκό. Πρέπει να σκεφτούμε, νομίζω ακόμα πιο καινοτόμα από ό,τι σκεφτόμαστε μέχρι τώρα. Και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Μέιστατ που υιοθετεί στην πραγματικότητα μια ειλικρινή και έντιμη τραπεζική προσέγγιση. Δεν θα ήθελε βέβαια η τράπεζα να λάβει πολύ περισσότερους κινδύνους, αλλά πρέπει, χρειάζεται να σκεφτούμε, να ψάξουμε να βρούμε και άλλες πρόσθετες απαντήσεις, γιατί όπως είπα οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι τεράστιες. Θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ τις εμπειρίες που διαθέτουν άλλοι για μια ε, υψηλότερη τόνωση των δημοσίων επενδύσεων, άλλους τρόπους για να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση. Εγώ θα επανέλθω στο θέμα των διαφόρων φόρων, για παράδειγμα επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά αυτή η πρόταση για τα καινοτόμα αυτά χρηματοδοτικά ε, μέσα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλαδή τα ε, ομόλογα για χρηματοδότηση ειδικών έργων, για χρηματοδότηση έργων, δεν θα αρκέσουν. Υποστηρίζω την ιδέα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα revolving funds, τα ανακυκλούμενα κεφάλαια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στις ε, δραστηριότητες της τράπεζας. Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα το Ευρωκοινοβούλιο και νομίζω ότι πρέπει να μπούμε και σε περισσότερο βάθος στην συζήτηση αυτή. Βεβαίως να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, αλλά να έχουμε σαφώς υπόψη μας ότι δεν επαρκούν αυτά για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 10 χρόνια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πρέπει να διακόψουμε για λίγο, διότι μου δήλωσαν από πλευρά του Επιτρόπου ότι πρέπει να αποχωρήσει. Λίγα λεπτά του μένουν. Τέλος πάντων, θα πει τώρα ε, ε, στο Επανιδίν και μετά θα συνεχίσουμε με τον Καρλ. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο, ο Επίτροπος Λεβαντόσκη, μία παρατήρηση επιτρέψτε μου να κάνω, ακούγοντας τις ανησυχίες που εκφράζεται, προέτους όταν γεννήθηκε ο μηχανισμός δημοσιονομικής σταθερότητας κυρίως στράφηκε γύρω από το θέμα της χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ως εγγύηση 60 δισεκατομμυρίων, 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα τουλάχιστον βλέπουμε ότι αυτό έχει ξεπεραστεί. Το ισοζύγιο πληρωμών θα παραμείνει, αλλά μπαίνουν τώρα διαρκείς μηχανισμοί βασισμένοι σε διακυβερνητική συνεργασία, χωρίς συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Θυμούμε τώρα τις ανησυχίες σας, θυμούμε και τις συζητήσεις μας, γιατί υπήρχε μέγας κίνδυνος εκείνη την εποχή. Τώρα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι διαφορετικό και νομίζω και αναγκαίο ε, δοθέντων των περιορισμών που αντιμετωπίζουμε και των κενών που έχουμε και στις υποδομές μεταφορών αλλά και στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και ούτω καθεξής την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την ενθάρρυνση μάλλον των ιδιωτικών επενδύσεων, είναι, συμφωνούμε με την αρχή που εξέφρασε ο πρόεδρος Μάιστατ, δηλαδή εξάντε κάπινγκ της συμμετοχής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. με οροφή για την, για την εξωτερική χρέωση το Ταμείο Εγγύσεων είναι μονάχα στη στάξη του 9%. και όχι το ποσό που δανείζει ε, ε, η Τράπεζα Επενδύσεων σε τρίτες χώρες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο κίνδυνα, κίνδυνοι απώλειας κλπ. Αυτό, αυτό θα είναι και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού σε οποιοδήποτε νέο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ε, ε, αυτές είναι, ε, αντιλαμβάνομαι και τις ανησυχίες σας βέβαια για δημοκρατική νομοποίηση κλπ. Σας ευχαριστώ. Ja, nochmal herzlichen Dank, äh, dass Sie... Η Πρόεδρος Ιωτα Χάουξ, σας ευχαριστώ που ήλθατε. Κύριε Επίτροπε, Συνεχίζουμε με τον κύριο Χάγκλουντ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τον πρόεδρο Μάιστατ γιατί έχασα το πρώτο μέρος της παρεμβάσεως του, του γιατί ψήφιζα σε άλλη επιτροπή. Η ομάδα των φιλελευθέρων πάντως ε, τάσεται ε, θετικά απέναντι σε αυτήν την ε, ιδέα Έχουμε και εμείς παρόμοιες ιδέες και αυτή που προτείνεται τώρα είναι πολύ παρόμοια με τις δικές μας, άρα είμαστε, ε, συζητούμε θετικά τις ε, σχετικές εξελίξεις. Λίγα σύντομα σχόλια. Πρώτα σχετικά με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κ. Καλφίν και που είναι ε, σωστές με την έννοια ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας με το μέσον αυτό. Αλλά δεν είναι και αυτό το θέμα. Είναι ένα μέσον αυτό και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά μην αποδυναμώσουμε τους, ε, τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για τράπεζα επενδύσεων. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνει. Το μοντέλο αυτό που μας υποβάλλεται τώρα είναι ευφιέ και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Τράπεζα Επενδύσεων για να προσελκύσουμε κεφάλαια για χρηματοδότηση σημαντικών έργων. Η πολιτική διάσταση εν προκειμένου είναι βέβαια η κατανομή ε, των ε, κονδυλίων. Μιλούμε λοιπόν για σημαντικά έργα σημαντικού ενδιαφέροντος και το ερώτημα είναι πώς και ποιος και πού θα λάβει τις αποφάσεις σχετικά με την χρήση των μέσων αυτών που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές πολιτικές συζητήσεις ίσως και συγκρούσεις. Αυτό χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Γνωρίζουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει στη διαθεσή της τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν έχουμε πρόβλημα καθ' αυτό κανένας μας αλλά εάν χρησιμοποιήσει αυτά τα καινοτόμα μέσα, το ζήτημα είναι πώς θα γίνουν οι επιλογές, γιατί εδώ τα πράγματα μπορεί να πάρουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιες σκέψεις σχετικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα, θα, θα ενδιαφερόμουν να τις, να ακούσω. Πάντως, με δύο λόγια, είμαστε, στεκόμαστε θετικά απέναντι στην ε, πρωτοβουλία αυτή. Helga. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤΕ για την παρουσίαση. Σε γενικές γραμμές τάσσομαι υπέρ αυτού του μέσου των project bonds γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση είναι, έχει πολύ υψηλό κόστος, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ευρώπης και χρειαζόμαστε νέα και βιώσιμη επένδυση. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε νέα φιλόδοξα μέσα έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να επενδύσουμε. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις ελεγκτικής φύσης ποια είναι η πρόσμιξη, η αναλογία ε, δανείων και grants και χορηγή και επιδοτήσεων και επίσης πώς ε, ελέγχουμε αυτό αυτό τον μηχανισμό τη στιγμή που η ΕΤΕ δεν μπόρεσε να ελέγξει τα private equities μέχρι τούδε. Θα ήθελα λοιπόν μία απάντηση σε αυτό το δύο ερωτήματα. Ο Ρίτσαρντ, ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο για την παρουσίαση. Θα ήθελα να πω ότι και εμείς τασόμαστε υπέρ του εγχειρήματο του. Μίλησε για διευρωπαϊκή υποδομή ή διασυνοριακές επενδύσεις. Ίσως να μην υπάρχει ε, δέλεαρ για το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στα κράτη-μέλη, διότι το μέγεθος, διότι αυτό αφορά το μέγεθος επένδυσης ή τον εμπλεκόμενο κίνδυνο στην επένδυση αυτή. Βεβαίως θα υπάρχουν ε, project στήριξη τη στιγμή που υπάρχει μία μακροχρόνια αξία. Θα ήθελα όμως να κατανοήσω καλύτερα τη διαδικασία προστασίας των φορολογουμένων. Πώς αξιολογείται τα προγράμματα Δηλαδή, όπως είπε και ο συνάδελφος, πώς ε, θέτετε προτεραιότητες, γιατί δεν μπορείτε να τα υποστηρίξετε όλα. Πώς αξιολογείτε την ποιότητα και πώς δίνετε προτεραιότητες, πώς ιεραρχείτε τις επενδύσεις. Επίσης, πώς προστατεύετε τους φορολογούμενους από την έκθεση σε κίνδυνο και ιδιαίτερα σε κίνδυνο στο οποίο δεν πρέπει να εκτίθεται. Ε, νομίζω ότι ο κύριος Μάιστατ θα μπορούσε να απαντήσει, αλλά εμείς ορίζουμε τις προτεραιότητες ως πολιτικοί και μετά εκείνος βλέπει κατά πόσο μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες επενδύσεις. Διαφορετικά δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ, εξ ονόματος της ομάδας μου, να πω το εξής. Πάντα είχαμε ταχθεί υπέρ των Eurobonds και η πρόταση εδώ των project bonds είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Δεν μπορώ να αποτιμήσω, ίσως τα Eurobonds διαφέρουν, αλλά η ιδέα των project bonds είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Εμείς συζητούμε, θα καθορίσουμε τη θέση μας, αλλά καταρχήν νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση που αξίζει να υποστηριχθεί. Πρόκειται για νέα χρηματοδοτικά μέσα. Θέλω εδώ να θίξω και μια άλλη διάσταση που ίσως θα έπρεπε να λάβει κανείς υπόψη όταν σχεδιάζει νέα χρηματοδοτικά μέσα. Διάφοροι και επιτόπου μου έχουν εξηγήσει και έχουν επίσης επικρίνει πώς γίνεται το monitoring επιτόπου σε ορισμένες τουλάχιστον περιφέρειες γίνονται, υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων για, γίνεται δηλαδή ασκείται κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί την ε, εκτέλεση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μια άλλη διάσταση και τελευταία εν προκειμένου που θέλω να τονίσω είναι η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων λειτουργεί σε τρίτες χώρες σαν τράπεζα επενδύσεων και καμιά φορά και σε ανταγωνισμό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εμφανίζεται εκεί ως δωρήτρια ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας. Αναπτυξιακής, όχι ανθρωπιστικής καλύτερα. Έτσι λοιπόν η αναπτυξιακης βοηθειας αναπτυξιακης οχι ανθρωπιστικης υπονομεύει εν μέρη τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας δηλαδή. Ίσως χρειάζεται να βρεθούν κάποιοι νέοι τρόποι συνεργασίας και κάποιοι νέοι ορισμοί των χρηματοδοτικών μέσων. Η κυρία Τζαβέλα. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας πρέπει να σας πω ότι επί της αρχής είναι εξαιρετική η πρότασή σας. Και συμβάλλεται ουσιαστικά πολύ θετικά κατά αυτόν τον τρόπο στο όλο ιστορικό της πρότασης αυτής. Ο κύριος Ντελόρ ήταν αυτός ο οποίος αναφέρθηκε πρώτος στο Project Bond. Εγώ τότε εργαζόμουν στον βιωτικό τομέα. Παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς την πρόταση του Προέδρου Ντελόρ τότε, η οποία προτάθηκε μεν αλλά κάπου χάθηκε στην όλη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Εν μέσω δύσκολων καιρών βλέπουμε να εμφανίζεται πάλι η πρόταση αυτή. Επί της αρχής λοιπόν είναι ένα πολύ καλό μέσο, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα τα οποία απομένουν ανοιχτά. Μέσω του μέσου αυτού κινητοποιούμε θεσμικούς επενδυτές, όπως είπε ο κύριος Μάιστατ. Μπορούμε όμως να κινητοποιήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να είναι αναγκαστικά θεσμικοί επενδυτές. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη. Τα έργα αυτά ξεπερνάνε ουσιαστικά τα έργα αυτά τα οποία καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρόκειται για άλλα έργα διαφορετικά. Και ποιος να λαμβάνει την πρωτοβουλία για την πρόταση των έργων αυτών. Δηλαδή, σε μια σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα κάποιος έχει την κυριαρχία, αν θέλετε, του έργου αυτού. Ποιος είναι owner στην περίπτωση αυτή ποιος είναι ο επικεφαλής του έργου αυτού και ποια έχουμε κάποια εμπειρία με τα corporate bonds, βλέπετε εσείς κάποιες ομοιότητες πέρα από όλα αυτά, πέρα από τις ερωτήσεις αυτές, πιστεύω ότι πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ καλό καινοτόμο μέσο. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Πρόεδρε τώρα παρακαλώ προχωρήστε στις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θα ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Έγγελ. Ενδεχομένως τα ποσά αυτά να φαίνονται τεράστια. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επενδύσεων αυτών μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι αποδοτικές επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις ε, μεγάλες εταιρείες παραγωγής και διανομής ε, ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαγορές. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και ε, συμφωνώ ουσιαστικά με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κάλφιν, μέσω των Euro Project Bond στοχεύουμε συγκεκριμένα έργα. Έργα τα οποία βρίσκονται σε μια ενδιάμεση, αν θέλετε, κατηγορία. Πρόκειται για έργα τα οποία δημιουργούν τα απαραίτητα αυτά έσοδα προκειμένου να μπορούν να υποστηριχθούν από Euro Project Bonds. Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε έργα τα οποία θα πρέπει να είναι αποδοτικά αλλά από την άλλη είναι έργα τα οποία έχουν ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου, το οποίο δεν επιτρέπει μια υψηλή βαθμολόγηση προκειμένου να μπορούν να αγοραστούν τα ομόλογα αυτά από τους θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται κυρίως για ιδιωτικές όμως εταιρείες. Πρόκειται για συνταξιδοτικά ταμεία, πρόκειται για ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικού οργανισμού, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα, αλλά κυνηγούν και ένα κάποιο υψηλό επίπεδο. Επομένω, η ιδέα των Euro Project Bonds σε καμία περίπτωση δεν είναι πανάκια και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση όλων των έργων. Μπορεί όμω να χρηματοδοτηθούν κατά αυτόν τον τρόπο τα έργα τα οποία μπορούν αργότερα να οδηγήσουν σε μια κάποια χρηματοοικονομική αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, χρηματοδότηση τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων ή διοδίων, για παράδειγμα, σε κάποιους κεντρικούς άξονες. Να έρθω τώρα στην ερώτηση της κυρίας Τρούπελ, που είναι πολύ εύστοχη. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε έργα τα οποία έχουν ε, ένα κάποιο μέγεθος. Εμείς χρηματοδοτούμε ουσιαστικά μία εταιρεία η οποία μπορεί να είναι μεικτή, ιδιωτική, δημόσια. Πρόκειται για την, την εταιρεία αυτή που έχει την κυριότητα που αναλαμβάνει να κατασκευάσει το έργο. Η εταιρεία αυτή θα έχει βέβαια κάποιο κεφάλαιο. Εμείς, και όταν λέω εμείς ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουμε μία πρώτη πίστοση, συμβάλλουμε χρηματικά και στη συνέχεια έχουμε το άλλο τμήμα της επένδυσης το οποίο έρχεται μέσω των Euro Project Bond. Δεν μιλάμε για σταθερά συγκεκριμένα ποσά, πάντως μπορούμε να πούμε ότι ε, για ένα έργο 100 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό πούμε το κόστος του έργου, στην περίπτωση αυτή 20 εκατομμύρια πρέπει να είναι το κεφάλαιο που έχει η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο αυτό. Εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων περίπου 20 εκατομμύρια και αυτό θα επιτρέψει λογικά να τοποθετηθούν 60 εκατομμύρια από έναν θεσμικό επενδυτή στη συνέχεια. Πρόκειται λοιπόν για ένα σχήμα το οποίο βασίζεται στο Transing, δηλαδή στο ότι γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα, μετοχικό κεφάλαιο, κύριο χρέος και υπαγόμενο χρέος. Στο παράδειγμά μου αναφέρθηκα σε αυτό το subordinated debt, στο μεσαίο δηλαδή αυτό, στη μεσαία αυτή στρώση, στο υπαγόμενο χρέος, το οποίο μπορούμε εμείς να καταβάλουμε ως ποσό μέσω διαπραγματεύσεων που θα γίνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δεσμευτεί ότι θα εγγυηθεί το ποσό αυτό το επίπεδο των 10-15 εκατομμυρίων ευρώ ή μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει το πρώτο ποσό και τον υπολοιπόμενο κίνδυνο θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πάντως σε κάθε περίπτωση εξ αρχής θα γνωρίζουμε ποιο είναι το μέγιστο κόστος, η μέγιστη επίπτωση για τον κοινοτικό προπολογισμό. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί το κόστος να αποδειχθεί σαφώς χαμηλότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντως και εξ αρχής θα γνωρίζουμε ποιο είναι το νότο ποσό το οποίο καλούμαστε να καταβάλουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα έργα. Ο κύριος Άσφορτ μας ρώτησε πώς αξιολογούμε τα έργα. Εμείς χρησιμοποιούμε τα συνήθι μας κριτήρια, δηλαδή τρία συγκεκριμένα. Πρώτον, το έργο αυτό θα πρέπει να συμβάλλει στην πραγματοποίηση ενός στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν, χρηματοδοτούμε οποιοδήποτε έργο μεταφορών, για παράδειγμα. Χρηματοδοτούμε τα έργα αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν έργα προτεραιότητας. Αυτό ονομάζουμε εμείς eligibility, eligibility criteria, κριτήρια επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τεχνικά, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά κριτήρια, προκειμένου να δούμε αν το έργο αυτό είναι βιώσιμο. Αν το έργο αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία πόρων, ακριβώς για να καταφέρουμε να αποπληρώσουμε και το χρέος το οποίο θα συνάψουμε. Και τέλος, στο τέλος, θέλουμε να δούμε αν πληρούνται και κάποια κριτήρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Δηλαδή θα πρέπει οι ιδιώτες, οι υπεύθυνοι του έργου αυτού να πληρούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αν πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια, τότε στην περίπτωση αυτή μπορούμε να υποβάλουμε το έργο αυτό στην, στο Δυτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον καταλαβαίνετε ότι μέσω συναπόφαση θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε τη χρησιμοποίηση αυτού του συνδυασμένου κοινού χρηματοδοτικού μέσου. Τα χρήματα του, Ευρωπαίου, του φορολογούμενου χρησιμοποιούνται μέσω του κοινοτικού προπολογισμού για αυτή την πολύ περιορισμένη συμβολή με ένα συγκεκριμένο πλαφόν που παίρνει τη μορφή εγγύησης που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, τα χρήματα του Ευρωπαίου του φορολογούμενου δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση πέρα από τα όσα αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν τα πράγματα εξελιχθούν θετικά θα χρησιμοποιηθούν και λιγότερα χρήματα γιατί ε, η μέγιστη αυτή δέσμευση τελικά δεν θα χρησιμοποιηθεί γιατί δεν θα χρησιμοποιηθεί τόσο υψηλό ποσό, το ποσό αυτό που έχει δεσμευτεί δηλαδή εξ αρχής για την εγγύηση. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του monitoring, της παρακολούθησης, προφανώς θα πρέπει να παρακολουθούμε τα έργα αυτά. Καθότι πρόκειται όμως για μεγάλα έργα, και απαντάω τώρα και στην κυρία Τρούπελ, δεν υπάρχει κάποιος ε, ε, διαμεσολαβητής, ε, χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής. Όπω είχαμε πει και παλιότερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε φορά που πρέπει να περάσουμε από για διαμεσολαβητέ, τίθεται πάντα το ζήτημα του ελέγχου που μπορούμε να έχουμε όσον αφορά την τελική χρήση των πόρων. Σαφώ έχουμε σημειώσει πρόοδο για το ζήτημα αυτό, αλλά εκ της φύσης τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Κάθε φορά που μιλάμε για μεγάλα έργα, εμείς προχωρούμε σε μια άμεση χρηματοδότηση, χωρίς να περνάμε από διαμεσολαβητές. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε πολύ πιο άμεσα τη χρησιμοποίηση των πόρων. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν στις συμβάσεις που υπογράφουμε πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τις αναφορές που θα πρέπει να υποβάλλονται και όσον αφορά τον έλεγχο των πόρων που επενδύονται. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ κύριε βουλευτές. Η Πρόεδρος Χάουκ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να είναι πολύ σαφέστερα τα πράγματα για όλες και όλους μας. Υπάρχουν ακόμη ερωτήσεις για τον ε, Πρόεδρο κύριο Μάιστατ. Ράιμα Μπέγκε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα ευχαρίστως ότι και αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, προγράμματα σε θέματα έρευνας μικρών και μεσών επιχειρήσεων και μεταφορών που έχουν σχέση και με τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό τα βλέπετε αυτά ως θετικά και ταχθήκατε και υπέρ της ιδέας να αναπτυχθεί περισσότερο ο μηχανισμός αυτός. Βέβαια και τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι άπειρα. Επομένως εν ώψη και των εξελίξεων θα γίνουν συζητήσεις με ποιον τρόπο ενδεχομένως θα επεκταθούν και οι δραστηριότητες σε τρίτες χώρες της τραπέζης σας. Μιλήσαμε λίγο και για νούμερα σχετικά με επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών καθώς επίσης και μεταφοράς ενέργειας. Είπατε και δικαίως ότι εν μέρη θα τα αναλάβει αυτά η ιδιωτική οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας, αλλά υπάρχουν και τομείς όπου θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη το δημόσιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Ποιες διαστάσεις της περαιτέρω εμπλοκής σας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, ιδιαίτερα για τα δίκτυα ενέργειας και τις μεταφορές, θεωρείτε εσείς ως δυνατή από πλευρά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Δεν ε, μπορώ να καταλάβω. Μιλάμε για 3-3 ευρώ. Δηλαδή αυτό ξεφεύγει από τη δυνατότητα κατανόησης, τη δική μου δυνατότητα κατανόησης. Μιλάμε για ε, γεωργία, υποδομές ε, και για πολλούς άλλους τομείς. Το πρόγραμμα Jeremy λειτουργήσε πολύ καλά μέχρι τούδε. Γιατί δεν μπορούμε να επινοήσουμε ένα ανάλογο ε, σύστημα και για τον ε, αγροτικό προϋπολογισμό. Σήμερα μιλάμε για μια μεγάλη ανάγκη επενδύσεων στον ε, περιβαλλοντικό τομέα κυρίως. Ιδιαίτερα για να αυξήσουμε την παραγωγή, για να μπορέσουμε να ε, προβάλλουμε να, να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες ε, νέα δις ανθρώπων συνολικά. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ε, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με το Ζερεμί. Μπορούμε να το αποκαλέσουμε ιεριχό για να του προσδώσουμε και μία ευαγγελική διάσταση. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε και στο γεωργικό τομέα, διότι ο γεωργικός τομέας είναι ο μεγάλος χαμένος. Αυτό είναι μια λανθασμένη προσέγγιση κατά την άποψή μου, διότι η γεωργία στην Ευρώπη θα πρέπει να βρει έναν τρόπο κάλυψης. Υπάρχουν, ε, πολλές, ε, υπάρχουν πολλά μικροεπενδυτικά σχέδια τα οποία καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτό θα ικανοποιούσε τους πάντες εάν θα μπορούσαμε να ε, προσφύγουμε στις σωστές ε, δανειοδοτήσεις, αντί να ζητάμε επιδοτήσεις συνεχώς. Ιζαμπέλ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα στοιχεία και την εισήγησή σας. Θα ήθελα να επανέλθω σε μία απάντηση που δώσατε σε σχέση με αυτό το κοινό επενδυτικό σχέδιο, γιατί μιλήσατε για αποδοτικότητα, αλλά και για ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις συνάμα. Μιλήσατε για τα συνταξιοδοτικά σχήματα ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί δεν υπάρχει πάντα απόδοση, ιδιαίτερα αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν πρόκειται για ιδιωτικές ε, χρηματοδοτήσεις. Δεν υπάρχει μία ρήξη συμφερόντων εδώ και μέσα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μας δεν θα έπρεπε να το ξαναδούμε αυτό, διότι οι ιδιωτικέ χρηματοδοτήσεις θα μας κατευθύνουν. Ιδιαίτερα ως προς το δεύτερο τμήμα της ε, διετησίας μας δηλαδή όχι μόνο monitoring αλλά και σύγκρουση συμφερόντων και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των ιδιωτικών επενδύσεων διότι έχω πολλά ερωτηματικά ως προς τη λειτουργικότητα του σχήματος. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εγώ διαρωτήθηκα πώς θα γίνει η πολιτική αξιολόγηση των έργων. Ότι μετά θα πρέπει να γίνει βεβαίως και η χρηματοδοτική αξιολόγηση, αυτό είναι σαφές. Καλά, θα δούμε. Βέβαια θα χρειαστεί κάτι να σκεφτούμε. Γιώραν Φέρμ. Ευχαριστώ. Μόλις σκέφτηκα το εξής. Εξήτασα προκαιρού την έκθεση Βιμ Κοκ για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατικής Λισαβόνας. Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της αναλύσεώς του ήταν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση για παράδειγμα με τις ΗΠΑ αλλά και με άλλα μέρη του κόσμου είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε το, είχαμε το χαμηλότερο τότε επίπεδο επενδύσεων. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη τώρα. Ακόμα έχουν εμφανιστεί νέα νούμερα που δείχνουν ότι στις αρχές, μάλλον το 2000, είχαμε ένα επίπεδο δημοσίων επενδύσεων περίπου της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ. Το 2015 θα έχει φτάσει στο 1,5%. Πρόκειται για μια απίστευτη πτώση, μια καταστροφική πτώση ε, των επενδύσεων. Και ε, ε, εδώ είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο επενδύσεων. Ασφαλώ βεβαίω ποιοτικών επενδύσεων. Αλλά πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο. Οι χώρε μέλη δεν μπορούν λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών τη κατάσταση του χρέου του. Δεν θέλουν επίση ούτε να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν θέλουν να αυξηθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε πράγματι καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό είναι προφανέ. Το δικό μου πρόβλημα είναι πώ θα το πλασάρουμε. Πώ θα πλασάρουμε την ιδέα αυτή στι χώρε μέλη αλλά και στι αγορέ κάναμε την προσπάθεια με εκείνες τις κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απόλυτη αποτυχία. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τους πείσουμε. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ορισμένες χώρες μέλη λένε «Α, αυτός είναι απλώς ένας τρόπος να επεκταθεί από την πίσω πόρτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλουμε να επεκταθεί. Έχουμε και άλλα προβλήματα διαφάνειας ε, καθολικότητας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, υπευθυνότητα και ούτω καθεξής. Έχουμε και άλλους μηχανισμούς και εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που αναπτύσσονται και προτιμούμε βέβαια να υπάρχει η ευθύνη, η διαφάνεια και ούτω καθεξής. Άρα πώς λύνουμε τα προβλήματα αυτά και τι ρόλο θα χρειαστεί να παίξουν οι χώρες μέλη και ποιο, ποιο θα είναι το όφελος υπέρ των χωρών μελών. Μπορεί να μας πει δύο λόγια ο κ. Μάιστατ για το πώς θα πλασάρουμε το προϊόν αυτό και στις χώρες μέλη και στους υπουργούς οικονομικών τους. κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν έλαβα απάντηση στο ερώτημά μου. Τα έργα αυτά ξεπερνάνε ουσιαστικά, είναι πέρα από τα έργα εκείνα τα οποία θα καλυφθούν από τα διορθωτικά ταμεία. Γιατί το Περιφερειακό Ταμείο, τα Ταμεία Συνοχής, καλύπτουν δίκτυα. Και ε, είναι γνωστό ποια δίκτυα θα καλύψουν. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από τα project bonds. Θα έχουμε ένα συνδυασμό διαρθρωτικών ταμείων και project bonds. Ε, δεν απαντήσατε σε αυτό μου το ερώτημα, Πρόεδρε. Ε, με κάθε σεβασμό. Ευχαριστώ. Herr Präsident, Ihre Antwortrunde. Παρακαλώ απαντήστε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω στον κύριο Μπέγκ ότι ε, μιλάμε εδώ μόνο για έργα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των έργων αυτών και μέσω των project bonds βέβαια, αλλά πρόκειται για ένα περιορισμένο αριθμό έργων για τα project bonds. Κατά τα άλλα μπορούμε προφανώς να συνεχίσουμε με τα εφιστάμενα μέσα να χρηματοδοτούμε τα έργα υποδομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το προσωπικό που έχουμε, με τα μέσα που έχουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση των έργων. Έχουμε δείξει ότι είμαστε σε θέση να είμαστε αθεκτικοί ακόμα και στι συνθήκε κρίση. Έχουμε το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής για τα υπόλοιπα χρόνια, τα επόμενα χρόνια. Διαφορετικά βέβαια θα πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα αν κληθούμε να κάνουμε και πράγματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη δράση της στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τα απαραίτητα μέσα αυτή τη στιγμή. Κυρία Πόλσεν, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας για τη γεωργία, γιατί εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε καθόλου στο γεωργικό τομέα. Γιατί εφόσον υπάρχει μια κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο επέμβαση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η απάντηση που δίδεται συνήθω παραδοσιακά στο ερώτημα αυτό και δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Κυρία Τζεβέλα. Ναι, όντω θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία, όπω ήδη συμβαίνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε το πρόγραμμα 3G, Jasper. Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει διαρθρωτικά ταμεία μαζί με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το πρόγραμμα Jeremy, για παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το οποίο έχει ως στόχο να μετατρέψει τα διαρθρωτικά ταμεία σε μέσα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει και με το πρόγραμμα Jessica όσον αφορά την ε, ανοικοδόμηση των ε, αστικών κέντρων. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τον συνδυασμό πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πόρων από τα διορθωτικά ταμεία. Και η επέμβαση μάλιστα, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των Project Bonds θα μπορούσε ιδίω για ένα έργο το οποίο θα έχει εγκριθεί από τα δροτικά ταμεία. Η συμβολή λοιπόν αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να χρηματοδοτεί και αυτή από τα διαρθρωτικά ταμεία του εν λόγω κράτου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στο ενδεχόμενο αυτό και θα μπορούσαμε να είχαμε μια διαφορετική χρήση των δραστηριοτικών ταμείων. Πάλι εδώ πέρα θα είχαμε αυτό το φαινόμενο τη μόχλευση, του πολλαπλησιασμού, αν θέλετε, τη θετική επίπτωση που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Η κυρία Ντιογόν στη συνέχεια έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση όσον αφορά την ποιότητα των επενδύσεων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο είπα και εγώ ότι θα πρέπει τα εν λόγω έργα να συμβάλλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι θα πρέπει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας δώσουν σαφείς ενδείξεις, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αν το έργο βρει είναι στον κατάλογο αυτό των έργων που είχε επιλέξει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τότε προφανώς και εμείς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το έργο αυτό, ακριβώς επειδή εξυπηρετεί τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απαραίτητα πάντα τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία δεν έχουν μια άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση αν το έργο είναι επιλέξιμο. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε αν είναι μια αλφα ποιότητα στο έργο αυτό, αν έχει την απαραίτητη, το απαραίτητο επίπεδο ποιότητος. Και βέβαια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία θα αξιολογήσει το στοιχείο αυτό. Και αυτό ο σημαντικό ρόλο, αν θέλει, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο νέο αυτό σύστημα. Να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε ακριβώ την επενδυτική αυτή ποιότητα, δυνατότητα του εν λόγω έργου. Ακριβώ και θεωρούμε ότι είναι λογικό να το κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή είναι σε θέση να κάνει αυτού του είδου την αξιολόγηση. Ο έλεγχο τη ποιότητα θα γίνει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι από του θεσμικού επενδυτέ. Εν κατακλείδη, συμφωνώ απόλυτα. Μετά όσα είπε με απόλυτη αυτοπεποίθηση ο κύριος Φαμ, Όντω ισχύουν όλα αυτά για τη στρατηγική τη Λισαβόνα και ισχύει και για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ευρώπη, αν θέλει να κρατήσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο και καλύτερα στο μέλλον και ιδίω στην έρευνα, την ανάπτυξη, την κοινοτομία. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον μα. Και πρέπει να βρούμε τους απαραίτητους αυτούς τρόπους που θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο τέτοιου είδους επενδύσεις, μολονότι διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ποιες είναι οι προσδοκίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναμένουμε όχι μόνο να χρηματοδοτήσει, να συμβάλλει τη χρηματοδότηση και των έργων που θεωρούμε άξια χρηματοδότηση, αλλά θέλουμε να σας ζητήσουμε και συμβουλές για την διαφήμιση που θα κάνουμε για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες αυτές από τις χώρες μέλη, τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής, για να πιστούν οι κυβερνήσεις ότι είναι δηλαδή η σωστή αυτή η προσέγγιση. Τώρα, ο εισηγητής μας λαμβάνει τελευταίο τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Μάιστατ για την εισήγηση αυτή. Αυτό που ανακαλύψαμε στη συνεδριά της Επιτροπής ΣΥΡ είναι τα όρια του κοινοτικού προϋπολογισμού και την ε, μεγάλη, την ύψιστη ανάγκη από πλευράς διαφόρων γενικών διευθύνσεων να προβάλλουν νέα χρηματοδότηση για να προωθήσουν τις κοινοτικές πολιτικές. Καθίσταται σαφές ότι δεν αρκεί ο υπάρχον προϋπολογισμός για να καλύψει όλους τους τομείς δαπανών και γι' αυτό όλοι οι επίτροποι που παρήλασαν από την Επιτροπή μας τόνισαν την ανάγκη παρέμβαση στη ΕΤΕ, ιδιαίτερα ως προς αυτά τα καινοτόμα μέσα παρέμβασης και μετά τις παρεμβάσεις του κυρίου Μαϊστάτ και τις αντιδράσεις των συναδέλφων καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να δούμε πού ελοχεύει ο κίνδυνος, πού ελοχεύουν κίνδυνοι και πού υπάρχουν ευκαιρίες. Θα πρέπει να δούμε την ευθύνη μας μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των νέων δημοσιονομικών μέσων για να ορίσουμε εξάντε άντε τις ανάγκες. Επίσης, Μέχρι το τέλος των εργασιών της Επιτροπής μας, Επιτροπής ΣΥΡ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες δαπανών, δηλαδή τι δαπάνες σχετίζονται με αυτά τα νέα καινοτόμα μέσα. Και ως προς τα, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές για να δούμε κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει η ΕΤΕ ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των project bonds. Η ΕΤΕ μίλησε για συμμετοχή των, της τάξης των 800 δις, δηλαδή τα δύο τρίτα του ετησίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις πιστώσεις ε, δαπανών. Και εάν λάβουμε υπόψη και το, το στοιχείο πολλαπλασιασμού, μιλάμε για 1,5%. Βρισκόμαστε στο 1,2% και υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ του 1,2% και του 5%. Άρα τα project bonds θα έχουν υψηλή συμμετοχή. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος. πολύ επέμειναν σε αυτό, το είπε και ο Επίτροπος, και θα πρέπει να δούμε και την συμμετοχή των δημοσιονομικών αρχών του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον ορισμό των σχεδίων και την έγκρισή τους. Η ΕΤΕ θα καθορίσει το πλαίσιο αλλά μιλάμε για ε, τον κοινοτικό προϋπολογισμό που θα λειτουργήσει ως εγγυητής. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε κατά τους επόμενους μήνες. Επίσης, ως προς την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων, θα πρέπει να αρκεστούμε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και των νέων στρατηγικών της Λισαβόνας. Θα πρέπει να μιλάμε για βιώσιμα σχέδια, δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουμε να καταβάλουμε το αντίτιμο αυτών των δανείων, στα πλαίσια δηλαδή αυτής της ε, δανειοδότησης, κάτι το οποίο υποστηρίζει το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια σύνοψη των παρεμβάσεων του κ. Μάιστατ και νομίζω ότι ως Επιτροπή ΣΥΡ ε, εγκρίνουμε, αξιολογούμε πολύ θετικά μάλλον αυτά τα σχέδια μέσα στα πλαίσια μίας ε, διάστασης που θα πρέπει να προσδώσουμε στο όλο εγχείρημα και χαιρόμαστε διότι η ΕΤΕ θα συμμετάσχει ενεργά έτσι ώστε να φτάσουμε σε βιώσιμες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ αγαπητέ Σαλβαδόρ. Νομίζω ότι σήμερα μπορέσαμε να λάβουμε πολλές απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις και μάλιστα απαντήσεις που θα μας βοηθήσουν στο περαιτέρω έργο μας. Βεβαίως πάντοτε εκπροσωπείται εδώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις συζητήσεις μας και παρακολουθεί τα όσα συζητούμε. Αλλά μάλιστα σήμερα ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρός της εδώ, ε, τον οποίον ευχαριστούμε ιδιαίτερος που ε, προσήλθε εδώ και απάντησε στις ερωτήσεις μας. Ελπίζω με αυτά τα Euro Project Bonds θα σημειώσουμε επιτυχία. Εγώ ήμουν και είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, διότι πραγματικά εφαρμόζει την κοινοτική μέθοδο, θέτοντας την πάντοτε στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ε, αν δεν έχουν οι συναδελφοί μου άλλες ερωτήσεις, σας ευχαριστώ που ήλθατε. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που άντεξαν μέχρι Τώρα, εάν δεν υπάρχει τίποτε άλλο για τα διάφορα, θα ευχηθώ σε όλους και όλους καλό σας βράδυ. Θα συναντηθούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και μάλιστα την Πέμπτη το πρωί. Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα μέχρι τότε.